Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι η πρώτη μας για το 2010. Ανεξάρτητα από το σημαντικό θέμα που έχουμε σήμερα να εξετάσουμε, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ευρωβουλευτές, όλους τους βοηθούς, όλους τους υπαλλήλους που μας βοηθούν στις εργασίες μας και όλους τους παρατηρητές που μας παρακολουθούν. Να ευχηθώ λοιπόν σε όλους σας καλή χρονιά για όλους σας και για τις οικογένειές σας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ακούσουμε τον υποψήφιο επίτροπο που έχει την ευθύνη των κοινωνικών υποθέσεων και της απασχόλησης, τον κύριο Λασλό Αντόρ, τον οποίο και καλωσορίζω εδώ για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας και ελπίζω ότι δεν θα είναι και τελευταία. Θέλω να επενθυμίσω τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε έτσι ώστε όλοι να γνωρίζετε πώς θα γίνουν τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο Επίτροπος έχει απαντήσει γραπτά στις γραπτές μας ερωτήσεις, στο γενικό πλαίσιο. Έχουν μοιραστεί στους συναδέρφους οι απαντήσεις του αυτές, σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση της γραμματείας έχει μοιραστεί στους ευρωβουλευτές είναι γεμάτη απαιτήσει ε, με κριτικό πνεύμα, έτσι ακριβώ όπως πρέπει να είναι και η δουλειά μας. Δέκα λεπτά λοιπόν θα δώσουμε καταρχήν στον υποψήφιο επίτροπο για να μας παρουσιάσει το έργο του και στη συνέχεια κάθε υπεύθυνο από πολιτική ομάδα στην Επιτροπή μας θα πάρει το λόγο. Μετά θα γίνει ε, ένας γύρος με ερωτήσεις βάσει του συστήματος DONT και στο τέλος θα δώσουμε το λόγο και στους συναδέρφους από την Επιτροπή Γυναικών και την Επιτροπή Πολιτισμού που βρίσκονται εδώ και εκείνες ε, μαζί μας και που συμμετέχουν σε αυτή την ακρόαση. Ένα λεπτό θα έχει ο κάθε ευρωβουλευτής, αυστηρά, ε? ένα λεπτό για να υποβάλει ερώτηση και δύο λεπτά θα έχει ο Επίτροπος για να απαντήσει στην κάθε μία από τις ερωτήσεις αυτές κάθε ερωτών μπορεί εφόσον το επιθυμεί να επανέλθει για το ίδιο όμως θέμα για να ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα για το οποίο έχει θέσει την αρχική του ερώτηση. Στο τέλος, μετά τις ερωτήσεις και των Επιτροπών Γυναικών 10 λεπτά και Πολιτισμού για, άλλα, για Συγγνώμη, διορθώνει πρόεδρος. 15 λεπτά θα έχει η Επιτροπή Γυναικών και 10 λεπτά η Επιτροπή Πολιτισμού. Μετά λοιπόν από αυτές τις ερωτήσεις θα μπορέσει να ολοκληρώσει ο Επίτροπος με μια πάλι μικρή παρουσίαση. Το κούρικο vitae του υποψηφίου Επιτρόπου έχει μοιραστεί όπως επίσης και η δήλωση συμφερόντων σας. Άρα είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Σας δίνω το λόγο για τα 10 λεπτά που έχετε στη διάθεσή σας για την αρχική σας παρέμβαση. Έχετε και ένα ρολόι μπροστά σας. Αν ξεπεράσετε το χρόνο σας, δυστυχώς θα αναγκαστώ να σας διακόψω. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. felelősséget is számomra. 15 éve idén, először... Φέτος, 15 χρόνια μετά, από την πρώτη επίσκεψη την οποία έκανα στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχοντας σε μια διεθνή διάσκεψη τότε γυρεύαμε μια απάντηση. Προσπαθούσαμε να δούμε ε, ποια είναι η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορεί να ενισχυθεί αυτή η κοινωνική διάσταση. Το ερώτημα αυτό παραμένει και σήμερα έγκυρο. Από την άλλη έχουμε προχωρήσει αρκετά, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα σε έναν τομέα ο οποίος πάντα με ενδιέφερε, και για κάποιον ο οποίος ε, θα έλεγα έχει βιώσει από την αρχή τις βαθύτατες αλλαγές που έγιναν στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και πάντα πίστευα στην ε, αναπόφευκτη κατά κάποιο τρόπο ε, ένταξη της χώρας μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη μεταμόρφωση και της δικής μου χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το καλύτερο. Η αναζήτηση της ευημερία και της προκοπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νομίζω ο στόχος τον οποίο πρέπει να έχει κάθε μέλος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συνεχίσω στα αγγλικά, λέει ο κύριος Σάντορ. Θα ήθελα <clears throat> να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την πολιτική ατζέντα της Ευρώπης. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη δική σας καθοδήγηση, συνεργασία και στήριξη. Για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και τις κοινωνικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειάζονται περίπλοκες προσπάθειες, αλλά είναι κάτι ιδιαίτερα στην, κατά τη διάρκεια της σημερινής κρίσης, κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια με κάθε ειλικρίνη αλλά και σκληρότητα η Ευρώπη αυτή τη στιγμή περνάει την πιο δύσκολη οικονομική κρίση της από την δεκαετία του 30. Έχουμε προβλήματα στον τομέα της απασχόλησης, υπάρχουν δείκτες έμβιας οι οποίοι αυξάνονται. Οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν ορισμένα προβλήματα τα οποία μεγενθύνονται, το ίδιο ισχύει και για τους νέους και για τους μεγαλύτερους ε, ηλικία εργαζομένους ε, τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με αναπηρίες, τους μετανάστες και αυτούς που ζουν σε στερημένες περιοχές. Η αηφορία λοιπόν του κοινωνικού μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβητείται. Γι' αυτό προτεραιότητά μου είναι να βρούμε μια έξοδο από την κρίση και να βγούμε πιο ενισχυμένοι από ό,τι στο παρελθόν. Απαιτείται άμεση δράση. Πρέπει να σταματήσουμε με μέτρα την απώλεια των θέσεων απασχόλησης. Υπάρχουν βέβαια και άλλες προκλήσεις όπως η γύρανση του πληθυσμού, οι νέες τεχνολογίες, οι κλιματολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές και η αηφορία των συνταξιοδοτικών συστημάτων μας και η διάρκεια τους στο μέλλον. Απαιτείται να αντιμετωπίσουμε σφαιρικά τα επόμενα δέκα χρόνια. Η στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η σωστή στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 θα δώσει τα μέσα και τις εταιρικές σχέσεις που απαιτούνται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους συναδέλφους μου ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια, να δώσουμε όλοι μαζί μια ισχυρότερη κοινωνική διάσταση. Μια Ευρώπη πιο δίκαιη μέσω ε, της δημιουργίας περισσότερων δυνατοτήτων απασχόλησης, μέσω ευκολότερης πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση, μέσω της καταπολέμησης των διακρίσεων στους χώρους εργασίας, μέσω της προσπάθειας προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, και μέσω της βελτίωσης των κοινωνικών υπηρεσιών. Όταν λέγω για μια Ευρώπη πιο αηφόρα, εννοώ την δυνατότητα της αγοράς εργασίας να προχωρήσει προς μια οικονομία πιο έξυπνη, με λιγότερες εκπομπές άνθρακα και να δημιουργεί τις λεγόμενες νέες θέσεις, τις πράσινες θέσεις εργασίας. να προσπαθήσουμε επίσης να βελτιώσουμε τις συνθήκες μέσα από τις οποίες ο εργαζόμενος θα αποκτά νέες δυνατότητες και θα έχει δυνατότητα συνεχούς πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση. Και φυσικά να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση μέσω ακριβώς της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου στην Ευρώπη, να ενθαρρύνουμε την κοινωνικά υπεύθυνη διαχείριση των αλλαγών, των σχέσεων μάλλον ανάμεσα στους εργαζομένους και στην εργοδοσία και να προχωρήσουμε επίσης και την ιδέα της εταιρικής ευθύνης. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να συνεργαστώ και με τους συναδέλφους μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους Αρμόδιους κατά τομέα το όραμα μιας πιο δίκαιης και πιο σωστής Ευρώπης είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πετύχουμε αν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας με έξυπνο και θαραλέο τρόπο. Έχουμε καταρχάς τα πολιτικά μέσα στη διάθεσή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση της διαβούλευσης και στο συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών. Μπορούμε να υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή με δεδομένα, με αναλύσεις. Έχουμε επίσης την δυνατότητα να εμπλακούμε και στον σφαιρικό κοινωνικό διάλογο, να προωθήσουμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς το εξωτερικό Δεύτερον, έχουμε τα νομοθετικά μέσα στη διάθεσή μας, στον χώρο της εργασίας και στους κοινωνικούς τομείς. Πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι νομοθετικές δυνατότητες, οι οδηγίες υπάρχουσες πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως και σωστά. Πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζομένους από κινδύνους στο χώρο εργασίας, πρέπει να προστατεύσουμε επίσης και τα συμφέροντα των εργαζομένων, η αδίποτε νομοθετική πρωτοβουλία απαιτεί, ε, που θα λυθεί μάλλον, απαιτεί ε, να υπάρξουν ε, μελέτες επιπτώσεων στον κοινωνικό τομέα, όπως ακριβώς η αναθεώρηση της οδηγίας για το ωράριο εργασίας. Το τρίτο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι το χρηματοδοτικό και αναφέρουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και το Progress. Έχουμε επίσης ξεκινήσει και κάνουμε τα πρώτα βήματα και για το Ταμείο Μικροχρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της σαν παράδειγμα να δίδει τα χρήματα τα οποία έχει στη διάθεσή της εκεί όπου χρειάζονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, απλοποιώντας τις διαδικασίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και στα πλαίσια της νέας πολιτικής συνοχής για το 2011 και μετά. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί κυρίως από την συνεργασία ανάμεσα στους ενδιαφερομένους. Το θέμα δεν είναι μόνο να στοχεύουμε σε νέες μορφές ανάπτυξης και νέες θέσεις εργασίας το θέμα είναι να βελτιώσουμε τη ζωή αυτών που είναι οι πιο ευάλωτοι όπως οι Ρωμά. Δεν θα πρέπει να τους εγκαταλείψουμε. Είναι ευθύνη για την κοινωνία, είναι θέμα αλληλεγγύης. Η επιτυχία σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με τα κράτη-μέλη και με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Τα επόμενα πέντε χρόνια σκοπεύω να εργαστώ στενά μαζί σας, να συνεργαστώ μαζί σας και αναφέρομαι στα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι το θεμέλιο θα έλεγα της δημοκρατίας στην Ένωση. Η καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας και του αποκλεισμού σημαίνει καταπολέμηση και διαφόρων μορφών διακρίσεων και αναφέρομαι εδώ στις προσπάθειες της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας των Φύλων όπως επίσης και τις προσπάθειες της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση. Θα αφιερωθώ με κάθε δυνατότητα που έχω στην προώθηση των στοιχείων αυτών που θα βοηθήσουν να προοδεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελπίζοντας να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα το χαρτοφυλάκιο το οποίο μου προορίζεται εφόσον μου δοθεί να ασχολείται με τόσο σημαντικά θέματα όπως οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι πολίτες, η υγεία τους και η ευημερία τους. Η οικονομική κρίση είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά μας δίνει και τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και να φτιάξουμε καλύτερες κοινωνίες. Έτσι βλέπω το χαρτοφυλάκιό μου. Αγαπητά μέλη, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Σύμφωνα λοιπόν με τη διαδικασία που έχουμε καθορίσει, θα περάσουμε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές. Η πρώτη παρέμβαση είναι εκ μέρους του ΕΛΚ από τον κύριο Σαμπόρη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, Έχουμε ένα αντίγραφο από τι απαντήσεις σας στις γραπτές μας ερωτήσεις και λέτε ότι μία από τις κύριες προτεραιότητές σα είναι η βελτίωση του επίπεδου απασχόλησης και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Επίσης, λέτε εκεί, ότι θα ξαναδείτε τις οδηγίες για την απασχόληση στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 και ότι θέλετε να υπάρξει συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί όμως, διότι αν θέλουμε συμφωνία με το Κοινοβούλιο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια της συναπόφασης. Το Φεβρουάριο όμως εσείς θα υποβάλλετε δήλωση για τις αρχές όσον αφορά τις νέες σας ιδέες. Κατά το παρελθόν όμως, εντάξει, ας πούμε ότι ό,τι έγινε, έγινε μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα θέλαμε εσείς να μας ενημερώνετε για κάθε καινούργιο στοιχείο που υπάρχει όσον αφορά στρατηγικές για την απασχόληση. Απάντηση. Το πρόγραμμα για το 2020 είναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα που έχει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με τον αξιότιμο Ευρωβουλευτή για το ότι η προετοιμασία είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά. Μιλάμε για τις επόμενες δεκαετίες, για την επόμενη δεκαετία συγκεκριμένα μέχρι το 2020, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι δουλειά θα κάνουμε και πρέπει επίσης να φροντίσουμε να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο στη δουλειά αυτή. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να μας βοηθήσει να έχουμε ανάκαμψη από την ε, παρούσα οικονομική κρίση. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αν δεν δούμε τα πράγματα και πιο μακροπρόθεσμα, έχω την πεποίθηση ότι υπάρχει ευρεία συνένεση στην Επιτροπή για το πόσο σημαντική είναι η διάσταση της απασχόλησης. Το ξέρουν αυτό όλοι. Εγώ θα βασιστώ σε εμπειρίες από το παρελθόν, θα εξετάσω τις πρακτικές που ακολουθήσαμε κατά το παρελθόν, το πρόγραμμα της Λισαβόνας, που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, και τι αποτελέσματα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Γιατί υπάρχουν. Βέβαια, υπό το φως της πρόσφατης οικονομικής κρίσης πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό πάντως να φροντίσουμε να εξυγχρονίσουμε τα πράγματα. Συμφωνώ πάντως μαζί σας για το ότι θα μπορέσουμε με τη βοήθειά σας να κάνουμε μεγάλα βήματα προς τα μπρος. Θέλετε να συμπληρώσετε την ερώτησή σας. Ναι. Χαίρομαι που ακούω τον υποψήφιο επίτροπο να λέει ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την προετοιμασία που έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά δεν μου απάντησε επί της ουσίας για την ερώτησή μου. Δηλαδή δεν άκουσα κανένα νέο στοιχείο όσον αφορά την πολιτική απασχόληση. Ούτε και ε, μου φαίνεται να είναι ξεκάθαρο όταν μιλάτε για μια συμφωνία επί αρχών, εσείς πώς θα το χειριστείτε το θέμα. Πριν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλει πρόγραμμα, δεν θα ήταν καλό να έρθετε εδώ πρώτα σε εμά πριν ε, δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα της Κομισιόν. Ο υποψήφιος Επίτροπος. Υπόσχομαι ότι θα φροντίσω να έχουμε ένα καλό πρόγραμμα με ενημερωμένα στοιχεία, πιο εξυγχρονισμένο και θέλω να ενθαρρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει περισσότερο ενεργό ρόλο και να συμμετάσχει περισσότερο. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε το πρόγραμμα βάσει των πρόσφατων αλλαγών, των πρόσφατων εξελίξεων απασχόληση, η διάσταση της απασχόλησης ε, πρώτα απ' όλα είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί για ολόκληρη την Ευρώπη και για όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Οι κύριοι στόχοι από πλευρά της απασχόλησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά που φτιάχνουμε προγράμματα, είτε πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος, Κάθε φορά πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις διαφροντικές αλλαγές και να φροντίζουμε η διάσταση της απασχόλησης να είναι ευρεία. Επόμενος, κύριο Σταβάλ, παρακαλώ. Α, συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Αλεξάνδρος Σάρκας έχει λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Άντορ, καλώς ήρθατε. Σήμερα ξεκινάμε σίγουρα ένα νέο στάδιο συνεργασίας. Και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διώξουμε ό,τι ανησυχίες υπάρχουν. Ανησυχίες που έχουμε εμείς ή που έχουν οι πολίτες και τις βάζουν στην ιστοσελίδα μας. Δύο κυρίως πράγματα. Πρώτον, η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Ξέρουμε το δικαστήριο, πώς έχει χειριστεί διάφορες περιπτώσεις. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα και με την ερμηνεία όχι μόνο με την εφαρμογή της οδηγίας, όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να πάψουν αυτές οι ανησυχίες από τον κόσμο. <clears throat> Και έπειτα, για την απασχόληση. Τον τελευταίο καιρό, ε, οι συνθήκες μάλλον εργασίας, ξέρουμε ότι είναι πράγματα τα οποία επηρεάζουν την υγεία, για παράδειγμα, των ε, πολιτών. Ο κύριος Μπαρόσο υποσχέθηκε αλλαγές. Εσείς μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα τι θα αλλάξει στο μέλλον η Κομισιόν όσον αφορά την οδηγία για την απόσπαση και για το χρόνο εργασίας, χρόνο απασχόλησης. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω την προσέγγιση μου για αυτά τα δύο σημαντικά θέματα και κυρίως όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων που αναφέρατε πρώτα. Η προέλευση της νομοθεσίας αυτής έρχεται από δύο πολύ σημαντικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι ότι θέλουμε να διευκολύνουμε την ε, μετακίνηση των εργαζομένων και δεύτερον προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το κύριο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και αναφερθήκατε κι εσείς στις αποφάσεις του δικαστηρίου, είναι λοιπόν η ερμηνεία που γίνεται σε αυτές τις δύο οδηγίες υπήρξαν δύσκολες περιπτώσεις. Και πολλές περιπτώσεις που μπορεί να μην συζητιώνται συχνά εδώ, αλλά που όντως δημιουργούν προβλήματα όταν κάποιοι αποσπασμένοι εργαζόμενοι μπορεί να καταλήξουν στη φυλακή, για παράδειγμα, ή τέλο πάντων έχουν κάποιες ε, διαμάχες με την κυβέρνηση τη χώρα στην οποία βρίσκονται, με τις αρχές της χώρας εκεί. θέλουμε κοινωνικό διάλογο και αξιολόγηση αντικτύπου για να ξέρουμε τις απόψεις όλων. Χρειάζεται σίγουρα μια νέα προσέγγιση. Όχι μόνο για αυτές, ίσως και για άλλα. Ενώ εδώ την οδηγία για τον χρόνο απασχόλησης, τον χρόνο εργασίας. Για τον χρόνο εργασίας επίσης, αυτή την οδηγία, είναι πολύ σημαντικό και εδώ να έχουμε μια αξιολόγηση κοινωνικού αντικτύπου και οι κοινωνικοί εταίροι να έχουν χρόνο στη διάθεσή τους να εξετάσουν το θέμα. Είμαι βέβαιος ότι και από τις δύο πλευρές θα γίνουν προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί κάποια συνένεση, να υπάρξει τουλάχιστον αμοιβαία κατανόηση. Πάντως καταλαβαίνετε ότι στην ε, Ευρώπη έχουμε πολλές διαφορές, υπάρχουν πολλά θα έλεγα κοινωνικά μοντέλα και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την επικουρικότητα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά τις προσδοκίες που μπορεί να έχουμε. Παρακαλώ κύριε Σαρκάς, ε, συμπληρωματική ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, ευτυχώς που τον Επίτροπο θα κρίνουμε σήμερα και όχι την Πρόεδρο, γιατί αν έπρεπε να κρίνουμε την Πρόεδρο, κάθε φορά που δίνετε το λόγο σε άλλον αντί για μένα, θα είχα υποψίες. Τέλο πάντων, αστείευομαι. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα τη κοινωνική αξιολόγηση. Είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε με τους ευρωβουλευτές ώστε η κοινωνική διάσταση και τα δικαιώματα των εργαζομένων να λυθούν υπόψη εξίσου όπως ε, αναφέρονται και ελευθερίε στην συνθήκη. Αυτή είναι η πρόθεσή μου, να συνεργαστώ μαζί σας, όντως. Και είμαι έτοιμος για κάθε περίπλοκο ζήτημα, αλλά και για απλά ζητήματα, να έρχομαι ξανά και ξανά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συζητάω ακόμα και τέτα τέτ με κάποιους από εσά αν θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους των φιλελεύθερων η κυρία Μαριάν Αρκίν. Καλησπέρα σας ε, κύριε υποψήφιε επίτροπε. Ε, δύο ερωτήσει έχω να κάνω. Πρώτον, όσον αφορά τη γραπτή σας απάντηση στην ερώτηση παριθμών 2, όπου μιλάτε για την όλο και μεγαλύτερη σημασία τη παγκοσμιοποίηση. Ε, και την όλο και μεγαλύτερη συνδυσία ανάμεσα στις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω λιγάκι να το αναλύσουμε αυτό. Αυτή η αδιαφυσβήτητη διασύνδεση αυτών των δύο πολιτικών, οικονομικής και κοινωνικής, ε, τι ακριβώς ε, προτείνεται σε αυτόν τον τομέα. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι για αυτούς που ε, φροντίζουν τις οικογένειες. Ένας μέχρι κάθε πέμπτος ε, έχει αρμοδιότητα για να ε, μεριμνήσει για τους γυρότερους πιο ηλικιωμένους ε, συγγενείς. Θέλω λοιπόν να μα πείτε τι ακριβώς προβλέπετε για αυτού και δεύτερον ποιες είναι, ποια είναι τα μειονεκτήματα που βιώνουν αυτοί, παραδείγματο χάρη την ευελιξία της ρυθμής εργασία. Κατανοώ βέβαια ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τα κράτη-μέλη. Όμως η Επιτροπή ε, προτίθεται να ε, ρυθμίσει αυτά τα θέματα όσων ε, φροντίζουν τους περισσότερου ηλικιωμένου. The impact of the globalization. Uh, we have to use uh... Κοιτάξτε, όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Ε, συστήθηκε το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ε, και οι ε, κανόνες αμφισβητήθηκαν σε κάποιες φορές. Νομίζω λοιπόν ότι μπορεί κανείς ε, να καταφύγει εκεί σε περίπτωση μετεγκαταστάσεων όταν προκύπτουν Σημαντικέ, μεγάλες, ε, εκτεταμένες απολύσεις ε, στα κράτη-μέλη. Τότε μπορεί κανεί να καταφύγει σε αυτό το ταμείο. Από την άλλη, θεωρώ η νέα κατεύθυνση που υπάρχει είναι να ε, ξεκινήσει ένας παγκόσμιος διάλογος σε διεθνές επίπεδο. Ε, λόγω της παγκοσμιοποίησης έχουμε τώρα τις ε, δομές της ομάδας των 20 όπου θα συμμετέχουν και οι Υπουργοί Εργασίας και αυτό θα γίνει για πρώτη φορά στην Ουάσιγκτον τον Απρίλιο. Νομίζω λοιπόν σε αυτό τον διάλογο σε διεθνές επίπεδο πρέπει να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε για να εκπροσωπήσουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και επίσης και να εκπροσωπήσουμε τι τις ευρωπαϊκές αξίες στον ε, κοινωνικό τομέα. To continue with the second question, the family carers uh, are definitely. Τώρα όσον αφορά όσους ε, φροντίζουν ε, τους περισσότερο ηλικιωμένους και το οικιακό προσωπικό, αυτό έχει ε, σχέση με το ότι υπάρχει γύρανση του πληθυσμού. Ε, στην Ευρώπη έχουμε πολίτες που γυράσκουν, γύρανση πληθυσμού. Ε, χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους ανθρώπους που τους φροντίζουν, άρα και περισσότερους θεσμούς. Και Βεβαίω πρέπει να μεριμνούμε για του ηλικιωμένου. Είναι σημαντικό αυτό να του προσφέρουμε υποστήριξη. Και πρέπει επίση το θέμα να το εξετάσουμε και από το πρίσμα τη των δυνατοτήτων των κυβερνήσεων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός είναι ένας ε, σωστός τρόπος για να προχωρήσει κανείς, δηλαδή να αναγνωρίσει κανείς ε, το έργο όσων ε, φροντίζουν τους ηλικιωμένους που μπορεί να είναι και συγγενείς αυτών. Διακόπτη πρόεδρος. Ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε. Είπατε, αναφερθήκατε στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Πρόσφατα αυτή η Επιτροπή έστειλε ε, μία επιστολή. Μία ερώτηση. Είσαστε στην τρίτη σας ερώτηση. Έχετε δικαίωμα για μία μόνο. Αναφέρθηκε σε αυτό ο Επίτροπος. Συμφωνώ μαζί σας, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, κατόπιν τούτου στη συλλογματική μου ερώτηση θα μιλήσω για όσους φροντίζουν τους ηλικιωμένους. Μιλήσατε ε, για την βιωσιμότητα ε, των ε, συνταξιδοτικών συστημάτων και για τη γέννηση του πληθυσμού. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συμπεριλάβετε όσου φροντίζουν για του ηλικιωμένου. Γιατί πολλοί εγκαταλείπουν τη δουλειά του και χάνουν τη σύνταξή του. Και αυτό είναι ένα τομέα με τον οποίο πρέπει να ασχοληθείτε όταν θα επιληφθείτε του συνταξιδοτικού. Αναμφισβήτητα. Κοιτάξτε, στην πράσινη βίβλο που σύντομα θα εκδοθεί, θα εξετάσουμε το θέμα και κάτω από το πρίσμα της σύνταξης. Και νομίζω ότι πράγματι ε, πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχει κάποια εμπειρία του να συμπεριλαμβάνονται, στο να συμπεριλαμβάνονται ε, άτομα μιας οικογένειας που φροντίζουν τους πιο ηλικιωμένους σε συνταξιωτικά συστήματα. Jean Lambert. Χαιρετίζουμε αυτά που είπατε για την διάσταση του φίλου στην απασχόληση. Χαιρόμαστε που έχουμε έναν επίτροπο ο οποίος ε, ενδιαφέρεται να ε, συμπεριληφθεί και δική του διεύθυνση σε όλα τα θέματα της ε, κοινωνικής πολιτικής γιατί μας, μας απασχολεί σιγά σιγά η διάβρωση των αρμοδιοτήτων σε αυτόν τον τομέα. Και υπάρχουν διάφορα παραδείγματα, υγεία, οικονομία, αλλά όπως και εσείς είπατε θα αναφερθώ στην κλιματική αλλαγή και στη βιώσιμη βιώσιμη ανάπτυξη που και εδώ υπάρχουν στόχοι για το 2020. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ε, σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στη νέα τεχνολογία αλλά και στο, περάσι, στο πέρασμα από την παλιά τεχνολογία σε περισσότερο αποτελεσματική. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν περιβαλλοντική συνείδηση. Μέχρι τώρα η πρωτοβουλία έχει αναλυφθεί από άλλα μέρη και μέλη της Κομισιόν, άλλους επιτρόπους, όχι από τον Επίτροπο Κοινωνικών Υποθέσεων. Πώς μπορείτε λοιπόν εσείς να παίξετε σημαντικό ρόλο μέσα στην Κομισιόν έτσι ώστε να γίνετε πρωτοπόρος για κάποια θέματα τα οποία σιγά σιγά μετακινούνται προς άλλα χαρτοφυλάκια. Κοιτάξτε, νομίζω πρώτα απ' όλα πρέπει να συστήσουμε μια καλή συνεργασία ανάμεσα στους επιτρόπους. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να συστήσουμε επίσημες ομάδες, αλλά να υπάρχει συνεργασία. Τώρα, στα θέματα που αναφέρατε εσείς, ε, η κυρία Χίλντεγκαρτ και ο κύριο Ποτότσνικ ε, σίγουρα ε, θα έχουν περισσότερε αρμοδιότητες. Με αυτού ε, πρέπει κυρίω να συνεργαστώ και από κοινού να αναζητήσουμε το τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα των πράσινων θέσεων εργασία και πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα καταφεύγοντα και στο κοινωνικό ταμείο. Βεβαίω, μπορούμε σίγουρα να βρούμε κάποια κονδύλια σε αυτό το χαρτοφυλάκιο τα οποία θα μας επιτρέψουν να στηρίξουμε την αλλαγή στην οποία αναφερθήκατε. Um, να επανέλθω λίγο σε αυτό που είπατε, όχι μόνο τους επίσημους τρόπους, αλλά είχαμε κάποιες ανεπίσημες ομάδες εργασίας στο παρελθόν. Θα προωθήσετε αυτή τη μορφή συνεργασίας ή άλλες πρωτοβουλίες. Και αν προωθήσετε τις ανεπίσημες ομάδες εργασίας. Τι διάσταση διαφάνειας θα υπάρχει, πώς θα ενημερωνόμεθα εμείς για το πότε θα συνεδριάσουν, με ποιους κτλ. Σας είπα ότι δεν θα είμαι απλά διαθέσιμος, αλλά όταν υπάρξει πρόοδος γύρω από το συγκεκριμένο τομέα θα σας ενημερώσω αμέσως και εσύ της άλλης θα είμαι τακτικά στη διάθεσή σας, θα είμαι παρόν γύρω από τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Για την ομάδα της αριστεράς, η κυρία Τσίμα. Καλημέρα. Φέτος είναι η χρονιά κατά της ε, Φτώχεια ε, και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το Κοινοβούλιο πέρυσι ενέκρινε μια έκθεση για την προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωση ε, και την καταπολέμηση της φτώχεια κυρίως των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλείται λοιπόν η Κομισιόν να καταθέσει μια ε, αναλυτική έκθεση για το κατά πόσον τα κοινωνικά συστήματα στα κράτη-μέλη μπορούν ε, να διασφαλίσουν ε, εισοδήματα πάνω από το όριο της ε, φτώχειας. Εξάλλου, καλέσαμε την Κομισιόν να εκπονήσει μία κοινή μέθοδο για τον καθορισμό του κατώτατου ορίου επιβίωσης ε, και είπαμε ότι θα πρέπει επιτέλους ε, να υπάρχει ε, μεγαλύτερη σύγκριση, μεγαλύτερη δυνατότητα σύγκρισης των δυνατοτήτων που έχουν σε διάφορα κράτη-μέλη, κυρίως για να προαχθεί η καλύτερη ποιότητα ζωής των παιδιών. Εσείς ως μελλοντικό υποψήφιος, τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε για να στηρίξετε αυτό το έτοιμά μας και να το εφαρμόσετε στην πράξη το συντομότερο δυνατόν. Νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη φετινή χρονιά. Η χρονιά αυτή πράγματι αφιερώνεται στην ε, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της φτώχειας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για αυτά τα θέματα που θίξατε που είναι φλέγοντα. Θεωρώ ότι η ε, φτώχεια των ε, παιδιών είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο θέμα. Ε, ένα παιδί σε ηλικία 4 ή 5 ετών δυστυχώς πρέπει να δεχθεί ότι κάποιος άλλος θα αποφασίσει για το μέλλον του και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο σε αυτή την τόσο μικρή ηλικία τα παιδιά να μην έχουν τη δέουσα προσοχή από την οικογένεια και από το κοινωνικό περιβάλλον. Και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το υπόλοιπο τη ζωή του διαγράφεται πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό λοιπόν που μπορεί να κάνει η Κομισιόν είναι να εκφράσει αυτές τις ε, απόψεις ε, με, μέσω της ε, ανοιχτής μεθόδου του συντονισμού και νομίζω πρέπει να συγκεντρώσουμε δεδομένα, να προσφέρουμε στα κράτη-μέλη αναλύσεις και να βοηθήσουμε όσους ε, πιστεύουμε ότι πράγματι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα. Αναμφίβολα έχουμε χρήσιμη εμπειρία για το θέμα αυτό και μέσω του ανοιχτού συντονισμού οφείλουμε να ε, προσπαθήσουμε να προβάλλουμε καλά παραδείγματα και επίσης οφείλουμε να διαδώσουμε τις ε, καλές πρακτικές και να πείσουμε τα κράτη-μέλη να θέσουν στόχους. Θεωρώ ότι η χάραξη πολιτικής ε, καθίσατε πολύ σοβαρή όταν τα ίδια κράτη-μέλη βάζουν στόχους ε, για τα ίδια και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενθαρρύνουμε. Ε, κυρία Τσίμερα, θέλετε συμπληρωματική ερώτηση. Κοιτάξτε, η δική μου ερώτηση ε, είχε κατά κύριο λόγο στόχο να μας πει η Κομισιόν ε, μέχρι ποιο βαθμού προτίθεται να συμβάλλει έτσι ώστε να καταλήξουμε από κοινού σε κοινωνικά κατώτατα όρια ή να θέλετε να εκπονήσουμε κριτήρια βάσει των οποίων θα καθίσταται σαφές πότε πρέπει να υπάρχει κοινωνικοπολιτική παρέμβαση. Εν ώψη του μακρύ χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, μία σειρά οργανώσεων επισήμαναν ότι ε, αυξάνεται η ενεργειακή φτώχεια και είναι επίγοντο να βρεθεί κάποια λύση. Υπάρχει ένας ολόκληρος ε, κατάλογος που περιλαμβάνει κριτήρια για τον αγώνα ε, κατά της ε, ενεργειακής φτώχειας. Εσείς τι θα κάνετε, θα ασχοληθείτε με αυτό και θα παροτρύνετε και τους υπόλοιπους συναδέλφους να πράξουν και αυτοί το ίδιο δεν έχω ακόμα μελετήσει το πώς ακριβώς συνδέεται η ενέργεια με τη φτώχεια, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά πιο σημαντικά ε, προβλήματα. Όπως είπατε και εσείς, το βασικότερο είναι να συμπεριληφθούν αυτά τα θέματα που είναι καινούρια, αλλά πιστεύω ότι σε πολλά κράτη-μέλη, σε πολλές ε, περιοχές υπάρχουν ε, σημαντικά προβλήματα με την απασχόληση, ε, τα σχολεία, ε, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες ε, βοήθεια της οικογένειας. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας ότι πρέπει πράγματι να επιληφθούμε αυτών των νέων θεμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέλμερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Αντόρ, εμείς στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών Ενδιαφερόμεθα ιδιαίτερα για τις αρνητικές επιπτώσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής στην ευελιξία της αγοράς εργασίας. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνουν την ευελιξία των εργαζομένων, αυξάνουν το κόστος της εργασίας. Όλες οι οδηγίες που έχει περάσει, που έχει περάσει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρνητικές. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυξάνοντας το κόστος της εργασίας αυξάνεται και η ανεργία. Τι θα κάνατε σαν Επίτροπος για να ελαφρύνετε τα βάρη αυτά, πώς θα ενισχύσετε την επικουρικότητα. Ανησυχούμε επίσης και για το ταμείο αυτό για την παγκοσμιοποίηση. Είναι πάρα πολύ μικρό και τα χρήματα που έχει στη διάθεσή του απορροφώνται από την διαχείρισή του και δεν βοηθούν περιοχές όπως η Ιρλανδία. σχετικά με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία γενικότερα. Το θέμα δεν είναι να επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις, το θέμα είναι να προστατεύσουμε τους εργαζομένους και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτά. Θυμίζω ότι σε πάρα πολλούς τομείς ε, της κοινωνικής πολιτικής υπάρχει η αρχή της επικουρικότητας η οποία κυριαρχεί και θα πρέπει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ε, να στρέφουν την προσοχή τους όταν χρειάζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Εγώ είμαι οικονομολόγος και δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι η εργασία είναι ένα απλό αγαθό Μπορούμε να μιλάμε για το κόστος και την τιμή του βιβλίου, του αυτοκινήτου ή δεν ξέρω και τι άλλο. Εκεί πράγματι υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης και φιλελεύθερης αντιμετώπισης. Αλλά τώρα μιλάμε όμως για την εργασία, μιλάμε για τα, τα εισοδήματα των εργαζομένων, τα εισοδήματα των οικογενειών και πρέπει να διαφοροποιήσουμε λίγο το κόστος της εργασίας από το κόστος των αγαθών γενικότερα. Σχετικά με το μέσο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης, είναι αλήθεια ότι είναι ένα πολύ πρόσφατο οικονομικό μέσο, ταμιακή διευκόλυνση θα έλεγα, και ίσως και να υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία να μην λειτουργούν με ικανοποιητικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά είναι μια θετική καινοτομία και βοήθησε αρκετά για να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι απολυθέντες εργαζόμενοι. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα αν το κόστος διαχείρισης και συμβούλων είναι υπερβολικό, πρόπονος θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα και θα ήθελα να το εξετάσω προσεκτικά πριν εκφέρω μια τελική άποψη. Ο κύριος Χέλμερ, ευχαριστώ κύριε Άντορ φαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται ότι αυξάνοντας τα δικαιώματα αυτών που εργάζονται ε, μειώνει κανείς τις δυνατότητες των ανέργων να βρουν θέσεις απασχόλησης. Στην ουσία εσείς είσαστε προκατελημένος και αρνείστε να δείτε τις προτεραιότητες της δυναμικής της αγοράς εργασίας. Εσείς ε, είσαστε εκδότης ενός ακροαριστερού ε, περιοδικού, είσαστε εναντίον του ΝΑΤΟ, εναντίον της ελεύθερης οικονομίας, ήσασταν και εναντίον των κριτηρίων του Μάστρη. Καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ευρωβουλευτών αμφισβητούν την ικανότητά σας για να καταλάβετε τη συγκεκριμένη θέση. Ε, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάσατε τις απόψεις μου είναι λίγο στρεβλωμένος θα έλεγα, για να μην πω ιδιαίτερο στρεβλωμένος. Οι απόψεις μου είναι γνωστές, τις ε, επαναλαμβάνω και τώρα αν θέλετε. Ήταν παραπλανητικά αυτά τα οποία που είπατε και δεν μπορώ σε 1,5 λεπτό να αντιμετωπίσω όλα τα θέματα τα οποία θέσατε προς συζήτηση. Ευχαριστούμε από του Ευρωπαίου για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, κυρία Μάρα Μπιτζότο. Είπατε ότι θα προσπαθήσετε έτσι ώστε οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες των εργαζομένων. Εγώ ανησυχώ για την έλλειψη στοιχείων από πλευρά σας σχετικά με την μετανάστευση ε, από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ανάγκη να τεθεί τροχοπέδι στην μετανάστευση ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίων που έχουν χάσει τις ε, θέσεις εργασίας τους. Το να κρατήσουμε ανοιχτές τις πόρτες σημαίνει ότι αγνοούμε ότι σε επίπεδο απασχόλησης δεν υπάρχουν θέσεις για όλους και θα οδηγηθούμε σε αναπόφευκτες κοινωνικές συγκρούσεις. Εδώ και λίγο καιρό ο κύριος Μπαρόσο σε συνάντηση είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις στην Ευρώπη, ας ελπίσουμε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν δίδεται απαντήσεις στα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Ο Επίτροπος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι η μετανάστευση είναι κάτι που πρέπει να εξετάζουμε σαν ένα περίπλοκο μεν ζήτημα, αλλά από την άλλη μεριά σφαιρικά. Στα πλαίσια δηλαδή της ε, παγκόσμιας οικονομίας και μάλιστα να μην το βλέπουμε σαν πρόβλημα, σαν πηγή Πολύ συχνά βλέπουμε ότι η μετανάστευση των ανθρώπων δημιουργεί πιο πλούσιες κοινωνίες. Οι μετανάστες μπορούν να προσφέρουν νέες δυνατότητες, νέες προπτικές και στην ιστορία της ανθρωπότητας η μετανάστευση ήταν και μάλιστα μερικές φορές, ε, κατά κάποιες περιόδους συχνά, πηγή εντάσεων. Όμως υπάρχει μια θετική πτυχή. Στις πρόσφατες εμπειρίες που έχουμε και μάλιστα στις χώρες που είχαν πιο φιλελεύθερα καθεστώτα μετανάστευσης υπήρχαν λιγότερες δυσκολίες. Η πρώτη, η δεύτερη γενιά δυσκολεύτηκαν περισσότερο βέβαια να ενταχθούν στις κοινωνίες και αυτό είναι κάτι που χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως, θα πρέπει να δείξω ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό, μια που είναι στο χαρτοφυλάκιό μου τώρα, αλλά όχι από την πλευρά του αποκλεισμού. Πρέπει να συνεργαστώ με την Επίτροπο Μάλστρομ και την Επίτροπο Ρέντινγκ για να δούμε την νομική πτυχή του θέματος και την κοινωνική πτυχή των ζητημάτων αυτά, ώστε να υπάρχει μια συνοχή στην αντιμετώπιση μας. συμπληρωματική ερώτηση. Αυτά που λέτε έχουν αρνητικές κοινωνικές, θα έλεγα, επιπτώσεις πολλοί προστατεύονται που υποφέρουν από την οικονομική κρίση, προστατεύονται μέσα στο οικογενειακό θα έλεγα περιβάλλον. Κοιτάξτε κυρία Μπιζότο, θέτετε μία ερώτηση και πρέπει να επανέλθετε στην ερώτηση στη δευτερολογία σας. Έχω μια άλλη ερώτηση λέει η κυρία Μπιζότο. Θα πρέπει εδώ ίσως με αφορμή την κρίση να δούμε τι τεράστια σημασία έχει η παραδοσιακή οικογένεια σε επίπεδο ουσιαστικό και ηθικό. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να ενισχύσετε την οικογένεια, μιας και έχει τεράστια σημασία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Ε, I ε, We ε, Ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε, πρέπει κατά τη γνώμη μου να το προσέξουμε αυτό. Το χαρτοφυλάκιο βραχυπρόθεσμα έχει λίγα μέσα για να στηρίξει τις οικογένειες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών και να τις ενθαρρύνουμε να δώσουν περισσότερη προσοχή στις ε, οικογένειες, μεγάλες οικογένειες. όπου τα παιδιά συχνά αντιμετωπίζουν δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις. Ωραία, ολοκληρώσαμε με τους συντονιστές <clears throat> και τώρα περνάμε στα άλλα μέλη της Επιτροπής. Η πρώτη ερώτηση εκ μέρους του ΕΛΚ από την κυρία Σάρι Εσαγιά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Άντορ, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση χρειαζόμαστε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική για να ενισχύσουμε την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα των εταιριών. Την ευελιξία ασφάλεια. Πώς τη βλέπετε εσείς σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απαντώντας μου θα μπορούσατε να μου δώσετε και τον ορισμό της ευελιξίας ασφάλειας, γιατί ο καθένας καταλαβαίνει τον όρο αυτό, την έννοια αυτή τελώς διαφορετικά. Και εσείς είπατε ότι στηρίζετε την ευελιξία και ασφάλεια εφόσον σωστά ερμηνεύεται. Επότε λοιπόν ερμηνεύεται σωστά αυτή η έννοια, μπορείτε να μας πείτε. Η ευελιξία ασφάλεια είναι όντω ένας δύσκολος όρος. Στη γλώσσα μου μάλιστα είναι πολύ δύσκολο να τη μεταφράσουμε σωστά αυτή τη λέξη. Είναι συνδυασμός πάντως δύο ενιών, της ασφάλειας και της ευελιξίας. Ξεκινάει από το ότι αναγνωρίζουμε πως και τα δύο ε, χρειάζονται για να πετύχουμε τους ευρύτερους στόχους της απασχόλησης και της ε, κοινωνικής προστασίας. Συνεπώς, πρέπει τους στόχους αυτούς να τους δούμε ε, μαζί και αναμφίβολα δεν σημαίνει ότι είναι ευθύνη του ατόμου. Έχει να κάνει, έχει να κάνει με το πώς οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να έχουν καλύτερες επαφές ε, μεταξύ τους και με τους εργαζόμενους. Οπότε η βασική ιδέα είναι ότι πρέπει να έχουμε ευέλικτα συμβόλαια για τους εργαζόμενους, αλλά το άλλο σημαντικό είναι η διαβίω κατάρτιση προκειμένου να διευκολύνουμε την απόκτηση δεξιοτεχνήτων που χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και τις μεταβατικές περιόδους που θα προκύψουν στο μέλλον. Επίσης, είναι θέμα πολιτικών εργασίας και κοινωνικής προστασίας. Πώς μεταχειριζόμαστε τους άνεργους, τι επιδόματα, τι μεταχείριση τέλο πάντων έχουν στις διάφορες χώρες οι άνεργοι. Πάντως η ευελιξία ασφάλεια ως προσέγγιση έχει βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις τον πρόσφατο καιρό να αντιμετωπίσουν την κρίση. Υπάρχει διάλογος, υπάρχει μια, ένας διαφρωμένος διάλογος ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους εργοδότες, ανάλογα με τις καταστάσεις που προκύπτουν. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το ανθρώπινο δυναμικό, το ανθρώπινο κεφάλαιο, κάθε άλλο. Συμπληρωματική ερώτηση. Ανταγωνιστικότητα στις οικονομίες μας είναι κάτι πολύ σημαντικό, επειδή ακριβώς θέλουμε να ενισχύσουμε την απασχόληση. Οπότε, συμφωνείτε με τις χώρες που βασίζουν την προσέγγιση τους στα κριτήρια του Μάστερ, που πρέπει δηλαδή να τηρούν τα κριτήρια αυτά σταθερότητας. Συμφωνείτε με την γενική οικονομική προσέγγιση. Όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Συνοχή αναφερόμαστε σε εδαφική, οικονομική και κοινωνική. Και η οικονομική συνοχή είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή μας απασχολεί. Πώς εφαρμόζονται οι κοινέ αξίες, οι κοινέ αρχές δηλαδή. Έχει σημασία να κρατήσουμε τους κοινούς κανόνες και αρχές και να εφαρμόσουμε τους κανόνες αυτούς με υπεύθυνο τρόπο. Βλέποντας αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι τώρα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, διαπιστώνουμε ότι σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τις φορολογικές πολιτικές κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής της κρίσης. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό είναι καλό πράγμα να έχουμε κοινούς κανόνες και είναι καλό πράγμα η εφαρμογή των κανόνων να ανταποκρίνεται στις ε, κυρίαρχες συνθήκες. Σχετικά με τα κριτήρια του Μάστρεχτ και εδώ έχουμε θέμα ομοιομορφίας. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία ε, θα έλεγα αποφασίστηκαν εδώ περίπου και 20 χρόνια, πρέπει να δούμε αν είναι εφαρμόσιμα κατά από όλες τις συνθήκες ή μήπως όχι. Ευχαριστώ για τη σοσιαλιστική ομάδα ο κ. Κοφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Άντορ, είπατε ότι θέλετε να συνεισφέρετε με τις αρμοδιότητές σας στην πραγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γνωρίζετε επίσης και μας το υπενθυμίσατε άλλωστε ότι ένα από τα βασικά θέματα στα πλαίσια αυτής της δραματικής κρίσης την οποία βιώνει η Ευρώπη όπως και άλλες οικονομίες είναι η ανεργία, ιδιαίτερα η ανεργία μακράς διάρκειας, μια ανεργία πάρα πολύ σημαντική ποσοτικά, μια ανεργία η οποία από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να επιληθεί και να αντιμετωπιστεί επαρκώς σύντομα. Θεωρείται χρήσιμο οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα οι πολιτικές οι οποίες έχουν σαν στόχο την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης να μην υπόκεινται ή μάλλον να υπόκεινται σε ένα σύστημα ε, κινήτρων και κυρώσεων. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να βοηθήσει. Η ανεργία πράγματι είναι ένα σημαντικότατο πρόβλημα σήμερα και θα παραμείνει μαζί μας το φαινόμενο αυτό παρόλες τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε. Είναι αληθές. Πρέπει να προσπαθήσουμε όμως να αλλάξουμε λίγο τα χαρακτηριστικά αυτού του φαινομένου και να αλλάξουμε επίσης και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης και να μην εγκαταλείψουμε τον στόχο της πλήρους απασχόλησης που είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος και πρέπει να τον διατηρήσουμε. Νομίζω ότι το ιδανικό αυτό της πλήρους απασχόλησης πρέπει να παραμείνει και να βρούμε επίσης και τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξόδου από την κρίση και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση. Ιδιαίτερα σε χώρες όπου η απασχόληση ήταν προβληματική και πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Στη δεκαετία του 80 και του 90 η ανεργία ήταν σημαντικό χαρακτηριστικό των οικονομιών πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής, ε, ε, ορισμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είχαμε μακροπρόθεσμη ανεργία γύρω στο 10% σε πολλές χώρες. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τρόπους να μειώσουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό θα πρέπει να γίνει καταρχάς σε εθνικό επίπεδο βέβαια και ο συντονισμός των πολιτικών απασχόλησης ε, θα πρέπει να έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος. Υπάρχει μεγάλη διαφορετικότητα και ποικιλία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφοροποιούμε ε, τις χώρες μεταξύ τους, αλλά τονίζω ότι και οι τομείς μεταξύ τους πολλές φορές έχουν σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά για να πραγματοποιήσουμε την πλήρη απασχόληση απαιτείται μια συμπαγής και σταδιακή αύξηση της οικονομικής απόδοσης. Και αυτό απαιτεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις, έστω και μακροπρόθεσμα. Η κοινωνική συνοχή πάντως είναι το βασικό χαρακτηριστικό ή ανταγωνιστικού οικονομικού συστήματος. Εσείς έχετε λοιπόν κάποιες αρμοδιότητες οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με ε, μια κάποια συνεργασία και με άλλους επιτρόπους. Μήπως μπορεί να υπάρξει μία μορφή συνεργασίας ε, και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια αυτών των αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να προσφέρει και το Κοινοβούλιο στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων τους οποίους έχετε δέσει. Όπως είπα στην εισαγωγική μου παρέμβαση, θα πρέπει να, να εργαστώ στενά με τους επιτρόπους, τους υπεύθυνου για τη βιομηχανία και τις οικονομικές υποθέσεις και νομισματικές υποθέσεις. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας θα έλεγα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σύνολο τριών χαρτοφυλακίων και σχετικά ειδικότερα με την απασχόληση οι δυνατότητες τις οποίες έχω εγώ είναι σχετικά περιορισμένες. Μπορούμε να βοηθήσουμε την πλευρά της προσφοράς, αλλά σχετικά με την προσφορά της ζήτησης, αυτό εξαρτάται περισσότερο από άλλα χαρτοφυλάκια, από άλλους επιτρόπους. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστώ στενά μαζί τους, τον κύριο Ταγιάννη, τον κύριο Ρεν, να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις. Το θέμα δεν είναι να ονειρευόμεθα για ισχυρά ε, επίπεδα ποσοστών ανάπτυξης της οικονομίας 2 και 3% κατέτος, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπους συγκεκριμένους για να διευκολύνουμε τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Ευχαριστώ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κόσα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κοιτώντα ε, την οδηγία Α1208, διαπιστώνουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, διότι απασχολούν πάρα πολλούς ανθρώπους με αναπηρίες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε τα τρέχοντα επίπεδα απασχόλησης. Δυστυχώς όμως δεν τα καταφέρνουμε. Αν δείτε το 75% περικοπές που έχει γίνει για τη στήριξη ε, των μισθών, καταλαβαίνετε τι δυσκολία έχει δημιουργηθεί για τα άτομα αυτά. Θέλω να ξέρω, κύριο ε, Μπαρόσο, ο κύριο Μπαρνιέ, τι λένε. Μέχρι τώρα αυτό που έχουν πει είναι ότι είναι εθνικό ζήτημα. Εμεί όμω θέλουμε μια απάντηση. Νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο να ξαναδούμε τον κοινοτικό νόμο και να αλλάξουμε κάτι. Πείτε μας λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε για να προωθήσετε τη δημιουργία απασχόλησης σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την ε, αναθεώρηση της νομοθεσίας, την αλλαγή στην νομοθεσία, δεν το έχω προγραμματίσει αυτό ακόμα. Θα ήθελα να το ξανακοιτάξω όμως. Πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο. Ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, μεταξύ άλλων και τα άτομα με αναπηρίες, τέτοιες ομάδες λοιπόν να πλήττονται είτε σε κυβερνητικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων, πιο σκληρά εξαιτία αυτή τη κρίση. Είναι απαράδεκτο αυτό. Τώρα, σε τι βαθμό αυτό είναι κάτι που είναι αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με τους κανόνες για την καταπολέμηση των διακρίσεων, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει κάτι. Σίγουρα όμως πρέπει να συνεργαστούμε, να διαβουλευτούμε με τα κράτη-μέλη για τις πρακτικές που ακολουθούνται και εφόσον αυτές είναι σε βάρος των ευάλωτων ομάδων να σταματήσουν. Ευχαριστώ. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν 15 ε, εκατομμύρια άτομα που πλήττονται από αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουγγαρία και στις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να ξέρετε ότι 90% των ατόμων αυτών δεν έχουν δουλειά. Είναι άνεργοι. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει επιγόντως να αναλυθεί κάποια δράση, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κάποια στήριξη. Αν δεν έχουν στήριξη, δεν είναι σε θέση να απασχολήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Στη χώρα μου, την Ουγγαρία, υπάρχουν κανόνες για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες. Αν οι επιχειρήσεις δεν τηρούν αυτούς τους κανόνες, τους επιβάλλονται κυρώσεις. Και σε άλλες χώρες η δημιουργία απασχόλησης είναι προτερότητα. Λοιπόν, τελικά ποια λύση εσείς πιστεύετε ότι είναι προτιμότερη για να έχουμε απασχόληση. Eh, irány fontos függően attól, hogy eh, még az adott Κοιτάξτε, θεωρώ ότι οι λύσεις που αναφέρετε είναι πολύ σημαντικές ε, και εγώ ε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ε, μπορεί το κράτος μέλος να έχει κάποια εμπειρία και να ε, μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί την εμπειρία αυτή. Σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε να επιτύχουμε άλματα ε, στην πολιτική απασχόλησης, ούτε στην κοινωνική πολιτική. Και από κάθε κράτος μέλος μπορεί κανείς να περιμένει καλύτερες λύσεις και καλύτερη απόδοση. Αυτή λοιπόν, αυτό το χάσμα το οποίο ανέφερε αναφέρθηκε από εσάς. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο και υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες που υφίστανται αυτή τη στιγμή. Τώρα, εκ μέρους ε, των ε, σοσιαλιστών και ε, δημοκρατών, ο κύριος Φρεντερίκ Νταρντέν. Μήπως μπορείτε να μας δείξετε πού ακριβώς κάθεστε. Εδώ, εδώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, έλεγα ότι φέτος έχουμε το έτος ε, της ε, καταπολέμησης της φτώχειας. Ε, αυτό αναφέρθηκε και ως εκ τούτου οι στόχοι πρέπει να οριστούν σε όλα τα επίπεδα, κυρίως για να αποφευθούν οι ακραίες μορφές φτώχειας, έτσι ώστε να μην μεταφέρεται η φτώχεια από γενιά σε γενιά. Εσείς αναφέρατε ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερος συντονισμός, ανοιχτός συντονισμός για τα κοινωνικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα όμως, εσείς με τι τρόπο προτίθεστε να δραστηριοποιηθείτε στο θέμα των Αθηγάνων Ρωμά και ε, πώς ακριβώς αξιολογείτε τη δουλειά του προκατόχου σας ε, σε αυτόν τον τομέα. Σημαντική είναι και η φτώχεια των παιδιών. Παρότι υπήρξαν πάρα πολλές υποσχέσεις σε αυτόν τον τομέα, ο αγώνας ε, κατά αυτής της φτώχειας είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρξει αναφορά αυτής της φτώχειας των παιδιών, γιατί θεωρώ ότι αυτή πρέπει να είναι και μια μεγάλη προτεραιότητα. Μήπως πιστεύετε ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στη δική σας τη βοήθεια. Και θα ήθελα επίση να γνωρίζω, εσείς προτίθεστε να εκδώσετε μία ανακοίνωση που να αφορά γενικότερα στις καθολικές υπηρεσίες. Η ε, πρόεδρος. Ε. Για τους Ρωμά. To ε. Κοιτάξτε, ο ε, κύριος Σπίγκλα πέτυχε πάρα πολλά, κατόρθωσε να θέσει το θέμα των Ρωμά, των Αθηγάνων Ρωμά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, είναι λοιπόν προφανές ότι αυτό το θέμα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη δημοσιότητα. Προβάλλεται περισσότερο από ότι ε, πριν από τη διεύνηση. Βέβαια θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα για τα νέα κράτη, <laughs> για τα νεα κράτη-μέλη. Και ε, βέβαια το θέμα έχει επεκταθεί και στα άλλα γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση. Υπάρχει πολύ καλή εργασία των υπηρεσιών ε, με πολύ συντονισμένο τρόπο και αυτό οδήγησε ε, στο να είναι περισσότερο αποτελεσματική η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Θα συνεργαστούμε με την κυρία Ρέντινγκ και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προβάλλουμε περισσότερο τη δουλειά που γίνεται σε πολιτικό επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αναζητήσουμε μεγαλύτερους πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να στηρίξουμε τα προγράμματα των κρατών μελών για ε, μεγαλύτερη κοινωνική αφομοίωση. Ε, προηγουμένως αναφέρθηκα στην ε, παιδική φτώχεια και θέλω εδώ να πω και κάτι άλλο. Κοιτάξτε, σε χώρες όπως είναι η Ουγγαρία, παραδείγματος χάρη, από την οποία προέρχομαι εγώ, αυτά τα δύο προβλήματα επικαλύπτονται. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Βελγική Προεδρία κάνει τις προετοιμασίες της για την παιδική φτώχεια και ε, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. σχετικά με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πιο συγκεκριμένους στόχους σε επίπεδο του ελαχίστου εισοδήματος. Μπορούμε να συστήσουμε κάτι τέτοιο προς τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε την έννοια αυτή. Δεν είναι με ένα ερώτημα πάνω στο οποίο μπορώ να σας δώσω γρήγορα μια σύντομη απάντηση. Ξέρουμε ότι σε ορισμένες χώρες υπάρχει ένας ελάχιστος μισθός, μια ελάχιστη αμοιβή. Θα πρέπει να συγκρίνουμε τις εμπειρίες των χωρών αυτών, όπως επίσης και τις εμπειρίες χωρών οι οποίες δεν έχουν αντίστοιχες νομοθεσίες. Ξέρετε ότι το θέμα αυτό είναι θέμα που αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Πρέπει να σεβαστούμε την επικουρικότητα και θα πρέπει να εισάγουμε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα. Η αντιπρόεδρος μας, σε όνομα των φιλελευθέρων, η κυρία Λίνα, Ξέρουμε ότι τα συνδικάτα έχουν όλο και λιγότερα μέλη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί που δεν ε, είναι εγγεγραμμένοι σε συνδικάτα προστατεύονται κατάλληλα. Τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σαν δικαίωμα το να εγγραφεί ή να μην εργαστεί ε, κανείς στα πλαίσια ενός συνδικάτου. τα θέματα του ωραρίου εργασίας, σαν παράδειγμα. Οι δυνατότητες του opt-out που είχαν αποφασιστεί είναι κάτι το οποίο τα συνδικάτα θεωρούν ότι άπτονται των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Κάποιοι άλλοι θεωρούν το αντίθετο. Θα ήθελα εν πάση περιπτώσει την άποψή σας για τις υπερορίες σαν παράδειγμα. Πιστεύετε ότι είναι δικαίωμα των εργαζομένων ή όχι. σχετικά με τα opt-out. Υπάρχει οικονομική και νομισματική ένωση. Από τότε που υπάρχει αυτές οι εξαιρέσεις, γενικά θα έλεγα, δεν είναι η καλύτερη λύση. Πάντα θα πρέπει να προωθούμε κανόνες οι οποίοι θα πρέπει και να εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες. Εφόσον υπάρχει ένα θεμελιώδες εμπόδιο για την εφαρμογή μια τέτοια ρύθμιση σε μια χώρα, τότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πάντα η δυνατότητα του opt-out. Το opt-out πρέπει να είναι όμως προσωρινό. Πρέπει να έχουμε κατά νου και όσον αφορά την διάσταση του χρόνου και αυτό βέβαια δεν πρέπει είναι να επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε πρέπει να γίνεται σεβαστό. Αυτό που είναι σημαντικότερο είναι ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όσον αφορά τώρα στην ε, προαιρετική υπερορία, προαιρετικές υπερορίες. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν είμαι σίγουρος για το κατά πόσον μπορούμε εδώ να καταλήξουμε σε γενικευμένα συμπεράσματα. Εγώ πιστεύω ότι αν οι υπερορίες είναι εθελοντικές για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ε, πρέπει παρόλα αυτά να αναστηθούν τρόποι προστασίας των εργαζομένων και αυτό για λόγους υγείας και ασφάλειας. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αφήσουμε κάποιο περιθώριο για τα θέματα των προαιρετικών ε, υπεροριών, αλλά δεν θα πρέπει να ε, ξεπενιούνται και κάποια όρια. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή αναφέρει η έκθεση Κομισιόν ότι υπάρχουν 14 κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα της ε, αυτοεξαίρεσης. Και Πολλοί καταφεύγουν σε αυτή τη ρήτρα γιατί θέλουν να χρησιμοποιούν μια πολύ χαλαρή ερμηνεία της ε, εργασίας. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό αποτελεί κατάχρηση. Και μια άλλη ερώτηση που ακολουθεί έχει σχέση με αυτό το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία για το ωράριο εργασία. Πιστεύετε ότι η λίστα μπορούσε να είναι τα θέματα της υγείας να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά και να κατατεθεί μια άλλη οδηγία ε, για θέματα υγείας που θα εξετάζει αυτά και μόνο τα θέματα, τα θέματα της υγείας. Συμφωνώ μαζί σας ότι όταν θα επανέλθει η οδηγία για το χρόνο εργασίας πρέπει να έχουμε μια νέα προσέγγιση. Η τομεακή προσέγγιση μπορεί βέβαια να είναι κάποια λύση είναι όμως ε, σαφές ότι πρέπει να μάθουμε από τις ε, δυσκολίες ε, που προέκυψαν κατά το παρελθόν για να αναθεωρηθεί αυτή η οδικία. Το opting out, αυτή η αυτοεξαίρεση δεν είναι κατάχρηση, απλά εκφράζει διαφορετικές πραγματικότητες σε διαφορετικά κράτη-μέλη και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν θα, γίνει η... όταν θα ξανασυζητηθεί το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους του ΕΛΚ, το λόγο έχει τώρα η κυρία Ρεζίνα Μπαστός. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε υποψήφιε Επίτροπε. Αναφερθήκαμε στην ανεργία. Η ανεργία μεταξύ των νέων έχει αυξηθεί πολύ. 5 εκατομμύρια νέοι στην Ευρώπη είναι στην ανεργία. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μία τροπολογία που υπέβαλαν οι Πορτογάλοι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ που συμπεριλήφθηκε στον προπολογισμό για φέτος. Στην τροπολογία λοιπόν αυτή προτείνεται η δημιουργία ενός έρασμους πρώτης απασχόλησης που θυμίζει λίγο το πρόγραμμα έρασμος για τους νέους που κάνουν ανταλλαγέ μεταξύ τους. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Εσείς Κύριε Επίτροπε Αντόρ, γνωρίζετε το σχέδιο αυτό και εάν ναι, είστε διατεθειμένος να δημιουργήσετε αυτό το πρόγραμμα έρασμος για την πρώτη εργασία και με τι συγκεκριμένα μέτρα θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της ανεργίας των νέων και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης που απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους νέους. Δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Εγώ ξέρω μόνο το πρόγραμμα Ερασμό που χρησιμοποιείται στην ανώτατη εκπαίδευση. Όμως ευχαρίστω να μάθω και την πρόταση στην οποία αναφερθήκατε. Είναι μια καλή, ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Και μα ενδιαφέρουν ειδικέ προτάσεις. Η ανάληψη πρωτοβουλίας βέβαια είναι έργο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά. Πρέπει λοιπόν να το κοιτάξω, γιατί το θέμα της ανεργίας μεταξύ των νέων είναι όντως πολύ σοβαρό σε πολλές χώρες, όπου φτάνει μερικές φορές και το 35% και έχει επιδεινωθεί εξαιτία της κρίσης. Απειλείται η γενιά αυτή των νέων σαν την χαμένη γενιά. Αν λοιπόν υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν, όχι μόνο να αποφύγουμε τα χειρότερα, αλλά και να βρούμε καλές λύσεις, να ξέρετε ότι εγώ θα σας στηρίξω. Έχουμε το κοινωνικό ταμείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους ακριβώς σκοπούς. Ευχαριστώ, υποψηφία Επίτροπε, για τα όσα μας είπατε. Είναι κρίμα που δεν γνωρίζετε το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στον φετινό προπολογισμό. Ελπίζω να ενημερωθείτε σχετικά γρήγορα. Και έρχομαι και στη συμπληρωματική μου ερώτηση, πάντα για την ανεργία των νέων. Υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει καν να βρουν μια πρώτη δουλειά. Και τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να τους βοηθήσουν με επιδόματα ανεργίας γιατί ποτέ δεν έχουν δουλέψει. Τέτοιες περιπτώσεις πώς εσείς θα προτείνετε στα κράτη-μέλη να βοηθήσουν. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να στηρίξουμε προγράμματα των κρατών μελών που προσπαθούν να βρουν δουλειά για αυτούς τους ανθρώπους. Μερικές φορές χρειάζονται ειδικά προγράμματα στοχοθετημένα υπέρ αυτών των ανθρώπων. Σε ορισμένες χώρες μέλη έχουμε καλά παραδείγματα έχουμε θετικές εμπειρίες για το πώς αντιμετώπισαν το πρόβλημα κυρίως στην Ήπεθρο. Οι πόροι υπάρχουν. Αν ένα κράτος μέλος έχει μια καλή πρόταση, εμείς θα το στηρίξουμε και θα φροντίσουμε για τη χρηματοδότηση. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου του ΕΛΚ πάντα η κυρία Ντανούτα Χιασλόβγικα παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, στην παρέμβασή σας είπατε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την απασχόληση. Ελπίζω ότι ως Επίτροπος Αρμόδιος για την απασχόληση ε, ξέρετε ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε και αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε στο πρόσωπο του επόμενου Επιτρόπου είναι ένα όραμα. Ελπίζω να μπορέσετε να απαντήσετε στην απάντησή μου. Για να πετύχει η κοινωνική πολιτική χρειαζόμαστε μέσα. Ένα από τα μέσα που έχουμε είναι το κοινωνικό ταμείο. Ένα ταμείο το οποίο φτιάχτηκε πριν από μερικά χρόνια και καταρχήν κάθε φορά που έχουμε μια κρίση μπαίνει στο ειδόλιο. Εσείς πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ταμείο αυτό θέλετε το ταμείο αυτό να αποκλειστεί από τις πολιτικές συνοχής. Πώς θα χρησιμοποιηθεί επίσης το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ. Το Κοινωνικό Ταμείο αποτελεί μέρος και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της πολιτικής συνοχής. Θέλουμε οικονομική και κοινωνική συνοχή, περί αυτού πρόκειται. Θα παραμείνει έτσι. Τώρα τι δυνατότητες υπάρχουν για καλύτερη ρύθμιση. Αυτόνομη ρύθμιση του κοινωνικού ταμείου δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν καλό να αποσυνδεθεί από την συνοχή. Μπορεί βέβαια να εξυγχρονιστεί το ταμείο. Και είναι δυνατόν να υπάρξουν νέες καινοτόμες λύσεις. Όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο έχει ήδη γίνει, δηλαδή να δούμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ποιες είναι οι καλές εμπειρίες που υπάρχουν από εκεί. Έχουμε το Jasper, το Jessica, προγράμματα από τα οποία έχουμε καλές εμπειρίες για το πώς μπορούμε να βάλουμε μαζί διαφορετικές πηγές πόρων. Συχνά βάζουμε την οικονομία της αγοράς και άλλα τμήματα της οικονομίας τα χωρίζουμε. Όμως, ακόμα και αν ορισμένες δραστηριότητες κάποια τμήματα της οικονομίας χρειάζονται χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους, αυτοί που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο χρήμα πρέπει πάντα να έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στην ε, οικονομία αγοράς. Ευχαριστώ. Εγώ δεν βλέπω το όραμα στο πρόσωπό σας ακόμα. Θα ήθελα να ξέρω ότι από την πρώτη μέρα θα είσαστε σε θέση να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα. Εσείς μας δίνετε τεχνικές λύσεις χωρίς περιεχόμενο. Αυτό το χειρισμό που μας προτείνετε δεν τον βλέπω στην πράξη. Έπειτα με την αγορά εργασίας τι θα γίνει. Το Ταμείο στηρίζει λίγους μόνο, προκειμένου να ανέβει λιγάκι το επίπεδο ζωής τους, χωρίς όμως να εξυπηρετείτε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και ούτε και αγορά εργασίας βέβαια επωφελείται. Πώς θα το αλλάξετε αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι 9-10 εκατομμύρια άνθρωποι ε, χαίρουν στήριξη από το Κοινωνικό Ταμείο κάθε χρόνο. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Άρα το μέσο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ σας έδισα μια ένδειξη για το πώς μπορεί να γίνει ο εξυγχρονισμός του. Δεν θα γίνει σε μια μέρα, θα γίνει στην πρώτη περίοδο της Επιτροπής, η οποία θα ασχοληθεί με τη στρατηγική 2020 και σίγουρα η απασχόληση και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πράγματα που θα δούμε κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η κυρία Γιούτα Στάνιρουκ τώρα. Ε, κύριε Άννο, αξιότιμα κύριε Ανω, στις γραπτές σας απαντήσεις ε, λέτε ότι ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι η αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Κατά τη δική σας άποψη, τα κράτη-μέλη πώς πρέπει να ε, τακτοποιήσουν ε, τους προϋπολογισμούς τους και αυτό μπορεί να συνεπάγεται απώλεια θέσεων εργασίας αλλά και άλλες αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους. Ε, εκτός αυτού, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες λόγω της οικονομικής κρίσης προέκυψαν και ζημιές στο συνταξιδοτικό. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Η εμπειρία των ε, διαφόρων κρατών μελών ποικίλει ε, όσον αφορά τις επιπτώσεις ε, από την κρίση και αυτό εξαρτάται και από την δημοσιονομική τους κατάσταση και από την κατάσταση της οικονομίας σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτό αφορά κυρίως ε, τις ε, συντάξεις. Για μένα το θέμα που τίθεται είναι το πώς θα συνεργαστώ με τον κύριο Όλι Ρεν και τον κύριο Ταγιάννη ε, για τη στρατηγική εξόδου. Προφανώς αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, δεν είναι μια πρόκληση μόνο για μένα το πώς θα δρομολογήσω την απασχόληση στο πλαίσιο της στρατηγικής εξόδου. Είναι ένα θέμα συλλογικό και δεν είναι καταρχήν δικό μου θέμα ε, αφορά κυρίως ε, τον κύριο Ρεν. Εκείνος καλείται να ε, συντονίσει την μακροοικονομική πολιτική των κρατών μελών κυρίως των χωρών εκείνων όπου εμφανίζονται διωγγωμένα ελλείμματα. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστούμε όσον αφορά τι δικές μου αρμοδιότητες. Όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν εισαχθεί τα τελευταία δύο χρόνια για να αντιμετωπιστεί η κατάρρευση της οικονομίας και η αλματώδης αύξηση της ανεργίας, αυτά τα μέτρα θα πρέπει να αποσυρθούν με αργό ρυθμό και οι κυβερνήσεις ε, πρέπει να έχουν χρόνο και να αποκτήσουν και συμβουλές για το πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά έχοντας κυρίως ε, κατά νου το θέμα της απασχόλησης. Ε, το συνταξιωτικό σύστημα υποφέρει σε ορισμένες χώρες, όχι σε όλες. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν χώρες όπου η ε, συντάξεις μειώθηκαν όχι μόνο ως προς την ονομαστική τους αξία, αλλά και ως προς την πραγματική τους αξία. Και αυτό ε, ως συνέπεια της κρίσης. Θα έχετε και άλλη ευκαιρία για να απαντήσετε στη δεύτερη ερώτηση. Παρακαλώ. Η οποία είναι εξή κατά την προηγούμενη θητεία για να επανέλθουμε στο θέμα των συντάξεων δεν συμφωνήθηκε ε, η δυνατότητα μετάβασης ε, των συντάξεων, μάλλον το θέμα των διαδοχικών συντάξεων δεν ορίστηκε, δεν συμφωνήθηκε. Εσείς τι θα κάνετε. Κοιτάξτε, το θέμα των διαδοχικών συντάξεων είναι ένα θέμα ε, το οποίο δεν έχει σχέση με ένα, αλλά με περισσότερα θέματα που απασχολούν την κοινωνία και την αγορά εργασία. Η δυνατότητα μεταφοράς συντάξεων, η κινητικότητα είναι ένα θέμα, η γύρανση επίσης. Σύντομα λοιπόν θα υπάρξει μια νέα πράσινη βίβλος για τις ε, συντάξεις και αυτή η νέα βίβλος θα είναι το σημείο κίνησης για να επανέλθουμε στο θέμα και να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Θα προσφερθεί λοιπόν αυτή η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Αλλά πράγμα το θέμα των διαδοχικών συντάξεων είναι ένα θέμα που πρέπει να το επανεξετάσουμε. Εκ μέρους ε, των ε, Πρασίνων, επόμενη η κυρία Τουρούνεν έχοντας ε, κατά νου Σχετικά με την ανεργία των νέων, νομίζω ότι η απάντησή σας μέχρι τώρα δεν ήταν ιδιαίτερα πλήρης. Είναι μια τεράστια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σύντομα, θα χάσουμε μια ολόκληρη γενιά. Βέβαια τα θέματα γύρω από την απασχόληση αποφασίζονται κυρίως σε επίπεδο εθνικό. Τι μπορούμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε για να συντονίσουμε τις πολιτικές αυτές τις εθνικές. Τι μέτρα θα προτείνετε στα πλαίσια της νέας αυτής προσπάθειας που θέλετε να αναλάβετε. Τα μέτρα θα πρέπει να εγκριθούν προφανώς από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, γιατί όπως είπα ότι η εμπειρία αυτή μοιράζεται με διαφορετικό τρόπο σε όλες τις χώρες. Η ανεργία των νέων είναι ένα σοβαρό θέμα, όχι σε όλες τις χώρες, αλλά στη μεγάλη, σε μεγάλο αριθμό χωρών. Υπάρχει σαν σοβαρό θέμα και χειροτερεύει λόγω της οικονομικής κρίσης. Εμείς ε, δίδοντας τα δεδομένα που απαιτούνται, κάνοντας τις αναλύσεις που απαιτούνται, καταλήγοντας σε συστάσεις προς τις χώρες αυτές, ελπίζω να αντιμετωπίσουν καλύτερα το πρόβλημα. Το θέμα επίσης συνδέεται και με την εκπαίδευση και εδώ υπάρχει προφανώς ε, ένα έλλειμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων κατάρτισης. Δεν αντιμετωπίζουμε λοιπόν μόνο ε, συνοπτικά θα έλεγα κοινωνικά προβλήματα αλλά και μακροπρόθεσμα διαφροτικά προβλήματα γύρω από την υπόθεση αυτή. Και γι' αυτό θα στηρίξουμε τις χώρες οικονομικά όσο μπορούμε. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι έχετε στο νου σας. Εμείς ε, περιμένουμε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγάλη φαντασία και με κοινωνική συνείδηση. Να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που είναι μια νέα κατάσταση και πρέπει να την ε, αντιμετωπίσουμε. Περιμένω λοιπόν πιο συγκεκριμένες ιδέες. Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια ομάδα εργασίας ε, ειδικά για την απασχόληση των νέων. Να στοχεύσετε σε θέσεις εργασίας για τους νέους να βελτιώσετε τις ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας σε επίπεδο ποιοτικό. Θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις κύριε Αντόρ. I'm ready to consider all uh, these suggestions. I think this is, uh... Άκουσα αυτά που είπατε με ενδιαφέρον. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προσπαθήσουμε επίσης και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο να προχωρήσουμε. Ελπίζω να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την κατάλληλη ατζέντα. θα συζητηθεί το θέμα και με άλλους επιτρόπους, αλλά νομίζω ότι οι δυνατότητες τις οποίες αναφερθήκατε, όπως ε, μια ομάδα εργασίας η οποία να προβλέπει την αναζήτηση πιστώσεων για την εργασία των νέων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναζητήσουμε. Ο αντιπρόεδρος μας ο κύριος Τόμας Μάν, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Την 1η Μαΐου του 2011, σύντομα δηλαδή, τελειώνουν οι περιορισμοί για την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων. Στην Ευρώπη βρήκαμε ικανοποιητικές λύσεις που μας επέτρεψαν να είμαστε πολύ ευέλικτοι. Και από την άλλη, στα παλιά κράτη-μέλη υπήρξε μεγάλη αποδοχή για τη διεύνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, ε, ε, στις ε, νέες χώρες υπήρξαν αρκετές μεταβατικές ρυθμίσεις Υπήρξε λοιπόν διαφοροποίηση. Αυτά θα καταργηθούν ε, σε λιγότερο από ένα χρόνο ή λίγο πάνω από ένα χρόνο. Όμως αυτό δεν το έχουμε ε, καταστήσει σαφές, σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει ασάφεια. Και τι θα κάνει η Επιτροπή, τι θα κάνετε πολύ συγκεκριμένα για να μην έχουμε ένα σοκ προσαρμογής σε αγορέ εργασία που είναι έτσι και λιωτεταμένε. και για να αποφύγουμε ε, το ενδεχόμενο τη διαφυγής εγκεφάλων εργαζομένων, δηλαδή που θα μεταβούν σε χώρε με υψηλότερου ε, μισθού και αποζημιώσεις. Κοιτάξτε, πάντα πρόσεχα τις διάφορες μελέτες και αναλύσεις και υπάρχει φόβος για την κινητικότητα μέσα στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα υπήρχε. Ο κόσμος μετακινείται από τη μία χώρα στην άλλη για να βρει καλύτερη δουλειά ή καλύτερη πληρωμή. Αλλά είχε υπερεκτιμηθεί κάπως αυτό για την επόμενη περίοδο. Πρέπει να σταματήσουν ε, οι προσωρινοί διακανονισμοί με κάποιες χώρες μέλη και να έχουμε μια πλήρη ελευθερία διακίνησης για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αν υπάρχουν προβλήματα πρέπει να τα δούμε συγκεκριμένα. Προς το παρόν αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα πράγματα πάνε σύμφωνα με τις προσδοκίες μας και ότι εκεί που έρχονται πολίτες από τις νέες χώρες μέλη και πάνε στις παλιές, οι παλιές επωφελούνται πολύ από αυτούς. Ε, ήσασταν ε, λίγο σαφείς ε, κύριε Επιτροπή, ίσως μπορείτε να είστε λιγάκι περισσότερο σαφείς. Κοιτάξτε, ένα στοιχείο του περιορισμού της κινητικότητας σε πολλά κρατημέρη ήταν η λαθρέα εργασία, η οποία αφαιρεί από τους εργαζόμενους τα κοινωνικά τους δικαιώματα και επίσης αφαιρεί και από τα κράτη-μέλη φορολογικά έσοδα. Παραδείγματο χάρη, ο Επίτροπο κύριο Σπίγκλε είπε ότι θέλει να εξαναγκάσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν καλύτερους ε, κανόνες γιατί αυτό θεωρεί ότι αφαιρεί την κινητικότητα των ε, εργαζομένων. Εσείς λοιπόν τι θα κάνετε. Ε, πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα για να μην υπάρχουν περιορισμοί στην κινητικότητα των εργαζομένων. Δεν είμαι σίγουρος ε, για το κατά πόσον ε, κατάλαβα πλήρως την ερώτημα. Ίσως μιλήσετε πάρα πολύ γρήγορα για να μπορεί να μεταφραστεί. Εν πάση περιπτώσει, λόγω της ε, κινητικότητας ε, θα πρέπει να δούμε λιγάκι ε, την κοινωνική ασφάλεια, πώς ακριβώς ε, διασφαλίζεται, πώς προσφέρεται σε εργαζόμενους που μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία από την αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων πριν τελικά να λάβουμε κάποια νέα πρωτοβουλία σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρίζια Κονσάρη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, δουλεύουν τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει ανασφάλεια και φτώχεια. Πολλές φορές ακόμα και για αυτούς που έχουν δουλειά. Κύριε Αντόρ, μπορείτε παρακαλώ να μας ε, δώσετε συγκεκριμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην αγορά εργασίας για τους ανθρώπους αυτούς. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας όσον αφορά τη στρατηγική ευελιξία και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα των εργαζόμενων φτωχών δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την ευελιξία και ασφάλεια, πιστεύω έχει να κάνει περισσότερο με τις ευάλωτες θέσεις εργασίας. Σε πολλές χώρες έχουμε πολλούς που εργάζονται σε θέσεις εργασίας που δεν είναι σταθερές, που δεν έχουν εγγύησεις. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι δυνατότητες υπάρχουν για να μειώσουμε το κομμάτι αυτό της απασχόλησης που είναι οι ευάλωτες θέσεις εργασίας. Ορισμένες χώρες έχουν βρει κάποιες λύσεις. Πάντως το βέβαιο είναι ότι όσοι έχουν τέτοιες θέσεις εργασίας, ασταθείς, πρέπει να προστατευθούν και αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε με διάλογο με τα κράτη-μέλη. Uh, Ο κύριος Ρεν και εσείς αναφερθήκατε στην λεγόμενη έξυπνη πράσινη ανάπτυξη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι εννοείτε. Η έννοια αυτή προέρχεται από μια πρόθεση την οποία έχουμε να εξετάσουμε τις διαφορετικές αλλαγές οι οποίες προκαλούνται από τις κλιματολογικές συνέπειες και να τις δούμε με θετικό μάτι, να έχουμε ένα θετικό όραμα και να μην βλέπουμε τις συνέπειες αυτές σαν απλά μια αιτία και ένα επιπλέον άχθος, αλλά σαν μια δυνατότητα ανάπτυξης θέσεων απασχόλησης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τομείς όπως η ενέργεια με μικρές εκπομπές καυσερίων όπως επίσης και στις κατασκευές και στην οικοδομή, στις οικοδομικές δραστηριότητες. Αυτό βέβαια θα απαιτήσει κάποια αναπροσαρμογή του μεγέθους των δραστηριοτήτων οι οποίες ε, σε αυτή τη φάση είναι ιδιαίτερα αρνητικές σε επίπεδο εκπομπών. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και μέσω της απασχόλησης και μέσω της κατάρτισης. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ο κ. Λεγκαρίκ. Διαπιστώνει κανείς μια αύξηση εκ νέου των κερδών στα χρηματιστήρια από πλευρά των μεγάλων πιστοτικών ιδρυμάτων και ταυτόχρονα μας ανακοινώνονται πραγματικές καταστροφές σε επίπεδο απασχόλησης. Διερωτώ λοιπόν, θα συμφωνήσετε μαζί μου για να προσπαθήσουμε να οδηγηθούμε σε μια, μάλλον μια, να κάνουμε μια οδηγία η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στα επιχειρηματικά συμβούλια να μπλοκάρουν τα σχέδια των επιχειρήσεων για μετακινήσεις και κλεισίματα όταν έχουν κέρδη. Αντί να έχουμε μια οδηγία αύξησης ε, του χρόνου απασχόλησης, να έχουμε μια οδηγία που να δίνει κίνητρα στη μείωση του χρόνου απασχόλησης για να διευκολύνουμε τη μεγαλύτερη απασχόληση. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για οδηγίες. Πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για νέες πρωτοβουλίες και για νέες πρακτικές οι οποίες επεκτείνονται η εφαρμογή τους όλο και πιο πολύ. Οι επιχειρήσεις ενισχύονται και ενισχύονται γιατί η κρίση σε ορισμένους τομείς φαίνεται ότι έχει τερματιστεί και αυτό είναι θετικό. Θα πρέπει όμως να εφαρμόσουμε τις αρχές μας και να προσπαθήσουμε να οδηγηθούμε σε μία ανάκαμψη χωρίς να αγνοούμε την απασχόληση. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι η οικονομική ανάκαμψη χωρίς θέσεις απασχόλησης. Βλέπουμε λοιπόν τις βιομηχανίες ε, να έχουν πλέον κέρδη, αλλά η αύξηση αυτή των δραστηριοτήτων τους δεν οδηγεί στην πρόσληψη νέων εργαζομένων. Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο στο οποίο κάνω κριτική. Η κρίση δεν είναι για όλους. Κάποιοι κερδίζουν πολλά χρήματα. Κάποιοι έχουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια και απολύουν. Γι' αυτό ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ε, στις, ε, στα επιχειρηματικά συμβούλια για να μπλοκάρουν αυτά τα προγράμματα απολύσεων και να μειώσουν τον χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων αν χρειάζεται. Οι εμπειρίες με τα επιχειρηματικά συμβούλια μέχρι τώρα νομίζω ήταν σχετικά θετικές και κατά τη διάρκεια της κρίσης φάνηκε αυτό είναι ένα από τα μέσα τα οποία βοήθησαν να υπάρξει μια καλύτερη μορφή συνεργασίας και ανταπόκρισης στις προκλήσεις της κρίσης. Πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο μέσο και δεν μπορεί στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι περισσότερο. Ο κύριος Λάγιος Βόξ. συνειδητοποιείται ότι σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται η κατάσταση της δημόσιας διοίκησης με την παροχή υπηρεσιών. Αν δει κανείς την πολιτική στον τομέα της απασχόλησης και την πολιτική, την κοινωνική, ε, να υπάρχουν μερικές φορές διαπιστώνει κανείς ε, ε, να υπάρχουν ορισμένες αντιθέσεις. Είναι αλήθεια ότι η κοινωνική πολιτική θα μπορούσε να επηρεάσει για την προστασία των υπαρχουσών θέσεων απασχόλησης και να μην επιτρέψει την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Πώς βλέπετε εσείς ε, λίγο την ε, επίλυση αυτών των προβλημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε και το θέμα της παγκοσμιοποίησης, έχουμε το θέμα του Ταμείου για την αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά παρόλα αυτά θέσεις εργασίας δεν βλέπουμε να δημιουργούνται. Οπότε ε, μήπως τελικά τα κοινωνικά μέτρα αποδυναμώνουν την αγορά εργασίας και λειτουργούν εις βάρος της απασχόλησης. Εγώ θεωρώ ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών πολιτικών, των κοινωνικών πολιτικών δηλαδή και των πολιτικών απασχόλησης από την άλλη, ο συνδυασμός αυτός είναι ένας καλός συνδυασμός. Και οι πολιτικές αυτές συνήθως είναι θα έλεγα εναρμονισμένες μεταξύ τους. Είναι επίσης αλήθεια ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες ρυθμίσεις σχετικά με τις θέσεις απασχόλησης της υπάρχουσες και η κάλυψη ορισμένων ποιών εργαζομένων μπορεί να δημιουργήσει ορισμένα προβλήματα, αλλά αυτό είναι κάτι το επιμέρους και όχι κάτι το ε, οποίο να ισχύει ευρύτερα και μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι ένα κοινωνικό σύστημα προστασίας το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων δεν μπορεί παρά να βοηθήσει την απασχόληση. Και αυτό συμβαίνει γιατί ενθαρρύνεται η παραγωγικότητα μέσα από αυτά τα συστήματα προστασίας τα οποία βρίσκουν τους εργαζόμενους ικανοποιημένους. Η κοινωνική προστασία λοιπόν δεν είναι σε αντίθεση με την απασχόληση. Απαιτείται λοιπόν να υπάρχουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Αυτός θα πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος. Και οι κοινωνικοί κανόνες βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ε, να ε, οδηγούν συστηματικά σε μία μείωση του κόστους της εργασίας αλλά σε μία βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο με τη σειρά του θα προσφέρει προστιθέμενη αξία. Συμφωνώ με την πρώτη παρατήρησή σας λέγοντας ότι όταν αναφερόμεθα στην ποιότητα των θέσεων εργασίας δεν μπορούμε να αγνοήσουμε βέβαια το κόστος της εργασίας και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στην Ευρώπη επενδύσεων στην ποιότητα του εργατικού δυναμικού και αυτό δεν είναι κάτι το κακό βέβαια αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο να ισχύει για όλους. Αν δει κανεί την πολιτική στον τομέα της παιδείας, η κοινωνική πολιτική και η πολιτική της παιδείας είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Οι μη εξειδικευμένοι εργαζόμενοι αυτοί θίγονται κυρίως από ε, την έλλειψη των θέσεων εργασίας γιατί οι ανειδίκευτες θέσεις στην ουσία έχουν πάει όλες στην Κίνα. Συνεπώς ε, τα κοινωνικά μέσα και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση της ανεργίας μερικές φορές βρίσκονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Αναφερθήκατε... Αναφερθήκατε στους ανειδίκευτους εργαζόμενους και για τις θέσεις οι οποίες χάνονται προς την Κίνα και την Ινδία. Πράγματι εδώ θα χρειάζεται να υπάρξει μια κάποια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει δίδοντας δυνατότητες στους ανειδίκευτους να έχουν πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και σε μια δεύτερη φάση στις θέσεις απασχόλησης στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεπειών της αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας. Ο κύριος Μπεναμιάς ε, για τους φιλελευθέρους. Άκουσα ότι θέλετε να ξεκινήσετε ε, κάποιες επεξεργασίες σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες και τις ε, υπηρεσίες που παρέχουν προς τους εργαζομένους. Πρώτον, σχετικά με τις ε, λεγόμενες καθολικού συμφέροντος υπηρεσίες ή ενδιαφέροντος υπηρεσίες ή την κοινή ωφέλεια. Κυκλοφορεί έτσι και αλλιώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μνημόνιο και στοχεύεται επίσης και ε, η δημιουργία μιας οδηγίας η οποία να καθορίζει ακριβώς την έννοια και το νόημα των συγκεκριμένων αυτών υπηρεσιών. Όταν μιλάτε για κοινωνική οικονομία εννοείται το σύνολο <clears throat> των ε, εταίρων οι οποίοι έχουν εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα Μήπως θα πρέπει να ξεκινήσουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τα ταμεία τα οποία καλύπτουν ας πούμε τις επικουρικές συντάξεις. Αναφερθήκατε στις κοινοφιλείς υπηρεσίες και στην κοινωνική οικονομία. Νομίζω το κατάλληλο πλαίσιο για να εξετάσει κανείς τις κοινοφελείς υπηρεσίες από πλευρά της Κομισιόν είναι ένα πλαίσιο ποιότητας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κοινέ αρχές, αλλά πρέπει να δούμε και την ποικιλομορφία που επικρατεί στα κράτη-μέλη, τις διαφορές δηλαδή που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες που έχουν διαφορετικό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, για παράδειγμα. Πάντως σίγουρα μπορούμε να συνεργαστούμε υπέρ ενός πλαισίου ποιότητας. Έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση, την ποιότητα και τις καλές τιμές. Η κοινωνική οικονομία τώρα είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να κοιτάξω πάλι μέσα στην επόμενη περίοδο από καινούργια οπτική γωνία. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται μόνο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πρόκειται και για την στήριξη των κοινωνικών αξιών. Συνεργασία, τέτοια πράγματα πρέπει να δούμε στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας. Ίσως να μην ήμουν αρκετά ακριβής. Ξανά λοιπόν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας, κύριε Μπέναμιας, αν θέλετε να σας καταλάβει ο υποψήφιος Επίτροπος, να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα γιατί δεν σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Α, ευχαριστώ. Ναι, ωραία. Θα επιβραδύνω, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Νομίζω ότι περιμένουμε ορισμένοι ευρωβουλευτές από διάφορες υπηκότητες την οδηγία για τις υπηρεσίες ε, της Να ξέρουμε τι επιτρέπεται για τη χρηματοδότησή τους, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. Πολλοί συνάδελφοι που ήταν εδώ και στην προηγούμενη θητεία δούλεψαν με ψηφίσματα, με προτάσεις, οδηγίες και ο κύριος Σαρκάς και άλλοι. Έχει γίνει δηλαδή πολλή δουλειά. Εσείς όμως δεν μας είπατε τίποτα για αυτά. Εντάξει, τα τα αργά αυτή τη φορά κυρία Πρόεδρε, ρωτάει ο κύριος Μπενεμιάς. Ο υποψήφιος επίτροπος. Για το θέμα αυτό πρέπει να συνεργαστώ και με τον Αρμόδιο Επίτροπο για την εσωτερική αγορά. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να κοιτάξω την κοινωνική πτυχή και τους στόχους που ανέφερε και στην προηγούμενη απάντησή μου. Καλές τιμές δηλαδή, εύκολη πρόσβαση και ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Πάντως είναι κυρίως θέμα εσωτερικής αγοράς, πρέπει να ξέρετε. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του ΕΛΚ, το λόγο έχει η κυρία Πασκάλ Γκρουνέ. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, θα ήταν χρήσιμο η Επιτροπή να εξετάσει και τους νέους κινδύνους που προκύπτουν για την υγεία από την κατάσταση στους χώρους εργασίας. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα διάφορες μικές διαταραχές, οι οποίες ε, αποτελούν και το 2 τρίτο των επαγγελματικών ασθενειών ε, σε πολλές χώρες. Εσείς τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για τις οστεομυϊκές διαταραχές λοιπόν. Τι θα κάνετε στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ε, το θέμα αυτό για την περίοδο μέχρι το 2013. Ενώ η κοινοτική στρατηγική βρίσκεται στη μέση της φέτος, ε, θα υπάρξουν ανταλλαγέ κατά την Ισπανική Προεδρία. Ίσως λοιπόν πρέπει να υπάρξει κοινοτική πρωτοβουλία. Τι συγκεκριμένα μέτρα προτείνετε εσείς για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό στους χώρους εργασίας και πότε. Τι προθεσμίες βάζετε. ψήφιο επίτροπο, ο κ. Σαντόρ. Θέλω να επιταχύνω τι εργασίε με νέα νομοθεσία. Σίγουρα Υπάρχουν νέες μορφές ασθενειών, όπως οι οστομικές διαταραχές, Να ξέρετε ότι και εγώ, και εγώ είμαι θύμα. Όντω πρόκειται για νεοφανιζόμενους κινδύνους στους χώρους εργασίας που έχουν να κάνουν με τα γραφεία μας. Ξέρω επίσης και το κόστος. Δισεκατομμύρια χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Για να σας τα πω με δύο λόγια. Θα ήθελα μια σφιχτή προθεσμία. Ήδη φέτος πρέπει να προχωρήσουμε για ένα-δύο θέματα. Και χρειάζομαι τη στήριξη του Κοινοβουλίου βέβαια για να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα συγκεκριμένα μέτρα. Τι μέτρα θα μας προτείνετε. Αναφερθήκατε στις ασθένειες, το κόστος. Ναι, αλλά τι θα προτείνετε, τι μέτρα θα προτείνετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι πίσω από αυτές τις ασθένειες υπάρχουν ε, απολύσεις. Και οι απολύσεις δεν είναι μόνο για οικονομικούς λόγους, είναι και για τέτοιου λόγους. Και μετά οι εργαζόμενοι δεν ξαναβρίσκουν δουλειά. Τι θα κάνετε λοιπόν, έρευνα, στηρίξει στις επιχειρήσεις, έρευνα για τα μηχανήματα, για τα γραφεία, ναι. Μέτρα θέλω, συγκεκριμένα μέτρα, τι θα μας προτείνετε, ιδίως αν θέλετε σύντομα να προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα. Ο κύριος Σαντόρ. Η αρχική σας ερώτηση ήταν για τους εμφανιζόμενους κινδύνους στην υγεία από τους χώρους εργασίας. Και συγκεκριμένα αναφερθήκαμε στις οστομικές διαταραχές. Υπάρχει όμως και ένα θέμα που βρίσκεται επί και αυτό είναι το θέμα του καπνίσματος. Που είναι βέβαια πιο περίπλοκο θέμα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Οι διαφορές που υπάρχουν ε, στις διάφορες χώρες πρέπει να ληφθούν επίψη σοβαρά. Πάντως, το θέμα πρέπει να μελετηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εγώ αναφέρθηκα στις οστομικές διαταραχές. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Η κυρία Κίνγκα Κουιστόρα, τους Χριστιανοδημοκράτες. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω... Ε, Θέλω να προσπαθήσω εγώ να σας δείξω λίγο διαφορετικά αυτή την υπόθεση. Ε, λέτε ότι χρειαζόμαστε οριζόντια οδηγία για την πολιτική απασχόληση. Μετά από την κρίση, οι μακροοικονομικοί δείκτες έχουν βελτιωθεί κάπως, χωρίς όμως να βλέπουμε αντίστοιχη βελτίωση στο θέμα της απασχόλησης. Τι συγκεκριμένα μέτρα, τι απτά μέτρα, τι προγράμματα πρέπει να προωθηθούν για να έχουμε μακροοικονομικούς πόρους με αποτελέσματα στην απασχόληση. Εσείς ποιος θέλετε να βοηθηθεί. Πώς θα λάβουμε υπόψη μας τους ανθρώπους αυτούς που επιγόντως χρειάζονται βοήθεια. Για τις μικροοικονομικές πιστώσεις, λέει ο κ. Σαντόρ, πρέπει να σας πω ότι πάντα ήταν πολύ σημαντικό να μπουν στην ατζέντα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε κοντά στη λύση. Ο οικονομικός τομέας σε πολλές χώρες δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ανέργων και των χαμηλά αμοιβόμενων. Οπότε επιδεινώθηκε η κατάσταση. Εδώ αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε πώς μπορούν οι άνθρωποι να απασχοληθούν είτε σε μικρές επιχειρήσεις είτε να φτιάξουν οι ίδιοι μικρές επιχειρήσεις. Και για να το κάνουν αυτό βέβαια χρειάζονται πιστώσεις, χρηματοδότηση. Αυτή λοιπόν η μικροοικονομική ε, ενίσχυση μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Πρέπει να θεσμοθετηθούν τέτοιες μικροπιστώσεις και σε χώρες όπου δεν υπάρχουν ακόμα. Σε μερικές χώρες υπάρχουν. Και σίγουρα αποτελούν μια προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Και χαίρομαι που λέτε ότι θα στηρίξετε την ιδέα αυτή. Γιατί πιστεύω και εγώ ότι είμαστε στο τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ε, θέλω όμως να μου πείτε και ποιες κοινωνικές ομάδες θα επωφεληθούν διότι ακούσαμε νωρίτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, η Ρώμα που δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Αυτή η διευκόλυνση θα μπορούσε να βοηθήσει και αυτούς. Τα κράτη-μέλη όμως έχουν υιοθετήσει και άλλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η κρίση από την οποία πλήττονται περισσότερο αυτά τα, αυτές οι ευάλωτες ομάδες. Ο κύριος Σαντόρ, αν δούμε το θέμα των μικροπιστώσεων πάλι, Δεν μπορώ να σας δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση για το που πήγαν καλύτερα τα πράγματα. Η Γαλλία και η Ισπανία πάντως είναι δύο χώρες που έχουν τον θεσμό αυτό. Τώρα για τις χώρες όπου δεν υπάρχει, για παράδειγμα. Όμως η φτώχεια είναι μεγάλη. Αναγκάζονται με πολύ ψηλού στόχους να δανείζονται χρήματα οι άνθρωποι. Οπότε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτό είναι κάτι που είχε ξεκινήσει και πριν την κρίση. Η προσπάθεια δηλαδή για μικροπιστώσεις. Πάντως προς το παρόν η χρηματοδότηση έχει λιγάκι εξαντληθεί. Γι' αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να το ξαναδούμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ταβίτ Καζά τώρα έχει το λόγο εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκε ο υποψήφιος επίτροπος είναι σίγουρα πολύ σημαντικά. Η απάντηση όμως που μας έδωσε είναι πολύ γενική. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για την ανεργία των νέων, εδώ δεν βλέπουμε τι θα κάνει ή όταν μιλάμε για την ε, μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση και τις επιπτώσεις που έχει στην Ευρώπη. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά δεν βλέπω να καταλαβαίνετε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση στην Νότια Ευρώπη. Για την ένδια, εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Και κυρίως για την ένδια από την οποία πλήττονται τα παιδιά. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα. 17% των Ευρωπαίων πολιτών σήμερα ζουν σε χαμηλότερα επίπεδα ζωής, κάτω από το όριο της ένδυας. Τι θα κάνετε λοιπόν εσείς για να λύσετε αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα. Είναι πράγματι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μιλάω για τη φτώχεια που πλήττει τα παιδιά, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έτσι διαμαγείας μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα. Μπορούμε όμως να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε μέχρι τώρα. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τέτοια καυτά κοινωνικά προβλήματα. Φυσικά, εν μέσω κρίσης οικονομικής, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε τους ανθρώπους να σκεφτούν την κοινωνική διάσταση όταν οι ίδιοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Μιλήσαμε για τις μικροπιστώσεις πριν από λίγο. Είναι μία λύση, μία καινοτομία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε κάπως τις επιπτώσεις. Τα κρατημέλη πρέπει να βρουν νέες ευκαιρίες και εμείς μπορούμε με το Κοινωνικό Ταμείο να τους βοηθήσουμε. Αλλά βέβαια πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα από το κοινωνικό ταμείο θα δαπανηθούν σωστά και θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Δεν μπορώ όμως να σας δώσω μια ξεκάθαρη εικόνα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, ίσως να μην ήμουν αρκετά σαφή στην ερώτηση που έκανα. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς θα λύσετε αυτό το πρόβλημα. Τι θα προτείνετε δηλαδή εσείς ως Επίτροπος, εφόσον αναλάβετε τα καθήκοντά σας, τι μέτρα θα προτείνετε για να λυθεί αυτό το θέμα της ένδυας για τις μακροπιστές, μικροπιστώσεις. Πώς θα χρηματοδοτηθούν, ούτε αυτό μας το έχετε πει. Η ένδια είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Αυτό δεν έχει νόημα να συζητάμε γι' αυτό μωρέα λόγια. Δράσεις χρειάζονται, πράξεις. Οπότε ως Επίτροπος τι νέα δράση θα προτείνετε για να επιτευθούν τα επίπεδα τα οποία θα έπρεπε να είχαν επιτευχθεί ήδη για το 2010 και τα οποία δυστυχώς δεν θα δούμε. Για παράδειγμα, η κατάργηση του αποκλεισμού. Εσείς τι άποψη έχετε για τις προτάσεις που έχουν γίνει και τι νέες θα κάνετε ως νέος επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σαντόρ. Σωστά. Αν μπορώ να σας δώσω μια ολόκληρη απάντηση στο 1,5 λεπτό που έχω στη διάθεσή μου. Δύσκολο. Φυσικά πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε τις αιτίε της ένδυας. Να τις εντοπίσουμε και να τις καταπολεμήσουμε. Μιλάμε για το εισόδημα, μιλάμε για μέτρα στήριξης που θα μπορούσαμε ε, να θέσουμε σε εφαρμογή για τους ανθρώπους αυτούς. Πρέπει να κοιτάξουμε μακροπρόθεσμα και πάνω απ' όλα να δούμε τις πηγές. Γιατί ορισμένες ομάδες τη κοινωνία μας υποφέρουν από τον αποκλεισμό αυτό, ε, από την ένδια. Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε με κατάρτιση, με υγεία, πάρα πολλά, πάρα πολλά πράγματα. Αλλά πρώτα απ' όλα χρειάζονται τα αίτια της φτώχειας, τα αίτια του αποκλεισμού. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Χρειάζεται συνεργασία. Επίπεδο εκπαίδευση, υγεία, σα είπα, είναι δύο πράγματα από τα οποία πρέπει να ξεκινήσουμε και να προτείνουμε πολιτικές για αυτά. Και σε εθνικό επίπεδο βέβαια μπορούν να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Η κυρία Ελιζαμπέτ Μωράν Σαρτιέ έχει τώρα το λόγο. Κύριε Επίτροπε, είστε ερευνητή. Οι απαντήσεις σας μερικές φορές ε, ήταν επιφανειακές και δεν είχαν περιεχόμενο. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να εκλεγούμε από τους συμπολίτε μας και οι συμπολίτε μας περιμένουν αποτελεσματικές και συγκεκριμένες πολιτικές για την απασχόληση. Θα ήθελα λοιπόν για την απασχόληση να σας θέσω τέσσερις ερωτήσεις. Καταρχάς, ε, ο κανόνας είναι μία ερώτηση. Ναι, όλα αφορούν την απασχόληση, προφανώς. Γνωρίζω τον κανόνα. Πώς ε, να καταπολεμήσετε την απώλεια θέσεων απασχόλησης ανειδίκευτων. Πώς ε, θα βοηθήσετε για να προσαρμοστεί κανείς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πώς θα καταστήσουμε ε, το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση πιο αποτελεσματικό και πώς θα εντάξουμε 15 εκατομμύρια αναπήρων στις θέσεις εργασίας που θα τους οδηγήσουν στο εσωτερικό της κοινωνίας με τη σειρά της. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά θέματα και θα πρέπει να ειδωθούν από τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις. και διαφορετικού ε, τρόπου προβληματική θα έλεγε. Πρέπει να συνδυάσουμε τις, δίφτα, τις διαφορετικές πλευρές που έχει το χαρτοφυλακιό μου. Θυμίζω ότι σε επίπεδο παροχής κατάρτισης και εκπαίδευσης για απόκτηση δεξιοτήτων δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Το θέμα αυτό ήταν ήδη στην ε, ατζέντα της Λισαβόνας έχει υπάρξει κάποια πρόοδος και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Ταυτόχρονα έχουμε κάποια μέσα στη διάθεσή μας για να υποστηρίξουμε τις εθνικές πολιτικές εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και προγράμματα από πλευράς των κρατών μελών. Η απάντηση είναι γενική, αλλά οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες βρίσκονται στα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο. Τώρα για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχει διαφορετικούς στόχους. Από τη μία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των μεγάλων μετακινήσεων των εταιριών από τις χώρες της Ευρώπης σε άλλες χώρες του υπολείπου κόσμου και ταυτόχρονα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων σε επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και σωστής χρήσης των διαθεσίμων υποδομών που παρέχει η αγορά εργασίας σε κάθε μία χώρα ξεχωριστά. Νομίζω ότι δεν περάσαμε στην ουσία του προβλήματος. Έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα για να μπορέσουμε να εξελίξουμε τις υπάρχουσες πολιτικές και οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα μέσα από διαφορετικές μεθόδους. Πρέπει να πάρουμε πολιτικά μέτρα και ποιες είναι οι πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Το θέμα είναι πιο δύσκολο να τους ξαναφέρουμε στην αγορά εργασίας από το να τους κρατήσουμε στην αγορά εργασίας. Βλέπετε λοιπόν κάποια πολιτικά μέτρα τα οποία να διευκολύνουν την παραμονή των εργαζομένων. η απάντηση που σας έδωσα μπορεί να ακούγεται γενική, αλλά από την άλλη θα πρέπει όταν συζητάμε για θέματα ε, ευελιξίας και ασφάλειας να σκεφτούμε ότι η στόχος μας μακροπρόθεσμα είναι να κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα η απασχόληση. Θα επαναλάβω λοιπόν για μια ακόμη φορά τη μεγάλη σημασία που έχει η κατάρτιση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και να επαναλάβω την αιμονή μας στον κοινωνικό διάλογο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για να υπάρχει μια ευέλικτη προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στην παγκόσμια οικονομία. Τελευταία ερώτηση από πλευρά της δικής μας Επιτροπής. Ο Χιούς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η υγεία και η ασφάλεια είναι βασικό τμήμα του χαρτοφυλακίου σας και τον τελευταίο καιρό το έχουμε αγνοήσει ιδιαίτερα αυτό. Άκουσα αυτά που είπατε για τις μειοσκελετικές βλάβες και τις δυνατότητες ε, οι οποίες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε σχέση με τη χρήση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Πέραν αυτών, Έχετε κάποιες προτάσεις να κάνετε. Έχουν σκεφτεί τις συνέπειες εργασίας σε περιβάλλον με νέα στοιχεία τα οποία μπορεί να προκαλέσουν βλάβες. We dealt with that directive. So what would you have in mind as the content for a new action program? Όταν ας πούμε υπάρχει περιβάλλον εργασίας με νανοστοιχεία, έχουμε σκεφτεί για τις πιθανές βλάβες που μπορούν να προκληθούν. Το νέο πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να λάβει υπόψη να απαντάει ο υποψήφιος επίτροπος στα περισσότερα από τα προβλήματα στα οποία ήδη αναφερθήκατε. Το θέμα της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα Ένα θέμα είναι να λαμβάνουμε αμέσως υπόψη τις επιστημονικές πληροφορίες και τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε. Ε, για τα καπνό, σαν παράδειγμα, έχουμε ξεκάθαρες ε, επιστημονικές αντιλήψεις, ε, κρατούσες και πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε άμεσα όπου δεν το έχουμε κάνει. Σε σχέση με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα έτσι ώστε να καταλήξουμε κάπου και υπάρχουν και ακόμα πιο περίπλοκες καταστάσεις όπως κάποιες επικίνδυνες ουσίες σε μικρή πυκνότητα και εκεί δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία από πλευρά της επιστημονικής κοινότητας και δεν προβλέπεται να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στην ομοθεσία που προέβλεπεται. Πάντως έχετε προβλέψει ένα πρόγραμμα δράσης με συγκεκριμένο περιεχόμενο στο μέλλον. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να προτείνετε κάτι το ουσιώδες όμως το σύνολο των επιτρόπων της Επιτροπής με την ηγεσία του Μπαρόσο. Τι πρέπει να κάνετε για να πείσετε. δεν είναι μόνο το θέμα της προσωπικής εμπλοκής, είναι και το θέμα της ε, νομοθεσίας. Υπάρχουν, ξέρετε, συγκεκριμένες επεξεργασίες αυτή την εποχή σε θέματα που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο της εργασίας όταν συζητάμε τα ωράρια. Είναι θέμα λοιπόν όχι μόνο προσωπικής αντίληψης, αλλά υπάρχουν νομικές διαφορετικές ε, αντιλήψεις και το θέμα είναι ένα από τα πιο επίγοντα θα έλεγα στο συγκεκριμένο τομέα. Καλώς σας ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις θα τεθούν από τους συναδέλφους της Επιτροπής Γυναικών. Η πρώτη ερώτηση από πλευράς του Λαϊκού Κόμματος από, τη, από την κυρία Γιαρόκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφερθήκατε επανειλημμένα στις ε, πιο ευάλωτες ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνους που αντιμετωπίζουν πολλές μορφές ε, διακρίσεων, εκείνες ε, που πραγματικά με τεράστια δυσκολία βρίσκουν δουλειά, αντιμετωπίζουν ανεργία. Για μας, για την Επιτροπή των Γυναικών, αυτά είναι πολύ σημαντικά μηνύματα και θα θέλαμε επ' αυτού να συνεργαστούμε να γνωρίζουμε αυτό τον οδικό χάρτη για την ισότητα των δύο φύλων. Πάντως υπάρχει και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Δηλαδή όσοι ζουν ε, με το σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας, ε, τι ακριβώς προτίθεται να κάνετε για αυτούς. Ένας ε, από τους συναδέλφος, ο κύριος Σάφκοτσιτς, ο, ο Σλοβάκος, είπε ότι το 2005 η Ρωμά, που είναι μία από αυτές τις ομάδες για, στις οποίες αναφερθήκατε σήμερα εκτεταμένα, αυτοί εκμεταλλεύονται το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας ε, της χώρας τους. Υπάρχει μια τελείως διαφορετική δηλαδή άποψη από ό,τι ακούτε και θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Η δική του δηλαδή άποψη ότι οι Ρωμά εκμεταλλεύονται το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, αυτοί οι άνθρωποι ε, που είναι περιθωριακοί, κανείς δεν ασχολείται μαζί τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύετε ότι πραγματικά εκμεταλλεύονται το σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας. Κοιτάξτε, εγώ τους Αθήγανους Ρωμά τους αντιμετωπίζω ως μια ομάδα με δική της αξιοπρέπεια, τους σέβομαι. Υπάρχουν πέντε κράτη-μέλη όπου ζουν οι άνθρωποι αυτοί και αντιμετωπίζουν όχι μόνο διακρίσεις και προκαταλήψεις, αλλά δεν έχουν και πρόσβαση στην απασχόληση, στο σύστημα υγείας, ε, στην κατοικία και σε πάρα πολλά άλλα προβλήματα συμπεριλαμβανομένης και της ε, εκπαίδευσης. Ως ε, συνέπεια λοιπόν αυτών των ε, προβλημάτων και του αποκλεισμού τους, εκεί καταλήξαμε να αντιμετωπίζουμε τους Ρωμά με αυτόν τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και αυτό το που αναφέρατε, η άποψη αυτή σίγουρα δεν είναι δική μου και δεν την υιοθετώ. Θα πρέπει να μιλήσω με τον συνάδελφο υποψήφιο, επίτροπο, για το θέμα και πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε, να κάνουμε αναλύσεις πριν καταλήξουμε και πριν ε, καταρτήσουμε μια νέα στρατηγική προσέγγιση για τους Αθήγανους Ρωμά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το θέμα το έχω ήδη συζητήσει με την κυρία Ρέντινγκ, αλλά θέλω να το συζητήσω και με άλλους ε, υποψήφιους επιτρόπους αργότερα όταν θα οριστούμε υποψήφοι κυρίως με αυτόν που θα είναι αρμόδιος για θέματα υγείας για να μπορέσουμε να έχουμε κοινή γραμμή σε τόσο περίπλοκα θέματα. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να κάνω και μία ε, ερώτηση ε, εγώ είμαι Ρωμά σε αυτό το κοινοβούλιο και ο λόγος που το ρωτάω είναι, είναι πολύ σημαντικό τι είδου ε, μηνύματα περνάει η Κομισιόν όταν πρόκειται για αυτή την ομάδα την ε, τόσο μειονεκτούσα. Θεωρείται ότι μπορεί να υπάρχει ένας κύριος Μίστερ, ένας Μαροσεύκοβιτς, που πρώτα είναι αντιπρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά δεύτερον είναι αρμόδιος για τις διαθεσμικές σχέσεις και τη διοίκηση και είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να έχει τέτοιου είδους απόψεις. Και μέχρι ποιου βαθμού μπορείτε εσείς να κάνετε κάτι. Ε, μπορείτε άραγε να παίξετε ρόλο του καταλήτη στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με πάση περιπτώσει, πώς ακριβώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους απόψεις στην Επιτροπή. Ε, λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει πρώτα να μιλήσω με τους ε, συναδέλφους. Πιστεύω ότι εδώ το πιο σημαντικό θέμα είναι να επιβεβαιώσουμε ότι κατά τη δική μας άποψη Μιλάμε όχι για μία ευάλωτη, αλλά κατά πάσα πιθανότητα για την πλέον ευάλωτη ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να την προσέξουν τα κράτη-μέλη να ε, εκπονήσουν στοχευμένα προγράμματα που προωθούν την συμπερίληψή τους και την ενσωμάτωσή τους. Ε, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από ό,τι έγιναν κατά τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Σα συγχαίρω, σας έχω ακούσει και σας συγχαίρω για τη δουλειά σας μέχρι σήμερα και ε, συνάδελφος Κόβατς ε, υπέβαλε μια πολύ σημαντική έκθεση. Νομίζω λοιπόν ότι ήδη υπάρχει κάποιο υπόβαθρο που μπορεί να μας βοηθήσει στο να προάγουμε νέες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. Και θα ήθελα να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Σπίτλα ε, εξέτασε το θέμα κατά την προηγούμενη θητεία ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικός. Η κυρία Στρέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε υποψήφιε Υπέτροπε, εγώ είμαι η συγγήτρια για την αναθεώρηση της οδηγίας που έχει να κάνει με την προστασία των εργαζόμενων γυναικών, εγγύων ή ελεχώνων. Υπάρχουν πολλές χώρες μέλη που έχουν νομοθεσία όσον αφορά την άδεια πατρότητας. Δεν υπάρχει όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για ίση κατανομή των οικογενειακών βαρών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Να λοιπόν, κάτι που μπορεί να βοηθήσει και την ισότητα των δύο φύλων και να βοηθήσει να συμφιλιώσουν ε, οι γυναίκες στην οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν την οδηγία 92-82, την πρόταση δηλαδή για την άδεια πατρότητας, αν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε αυτήν η άδεια πατρότητας. Εγώ στηρίζω την ιδέα. Την ιδέα δηλαδή και οι άντρες να ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά, οι πατεράδες. Εγώ το έχω κάνει και ξέρω ότι πολύ συχνά η άδεια πατρότητας μπορεί να βοηθήσει. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να γίνει και κάτι το υποχρεωτικό. Πριν καταλήξουμε, πρέπει να δούμε τι ισχύει, τι καλά παραδείγματα έχουμε στις διάφορες χώρες μέλη και να δούμε πώς μπορούν αυτές να συνδυαστούν με τα κοινωνικά συστήματα και τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στις υπόλοιπες χώρες. Γιατί και πάλι αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην αρχή της επικουρικότητας και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών μελών. Σας ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε. Βγάζω το συμπέρασμα ότι είσαστε υπέρ της ύπαρξης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την άδεια πατρότητας. Θέλετε να συμπεριληφθεί στην οδηγία 9282 μια τέτοια πρόταση για την άδεια πατρότητας ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει άλλη πρωτοβουλία χωριστά και αν ναι, πότε θα αναλάβει η Επιτροπή μια τέτοια πρωτοβουλία για την άδεια πατρότητας θα πρέπει να εξετάσω περισσότερο σε βάθος το θέμα, να είσαστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω να βρω την καλύτερη προσέγγιση και την καλύτερη χρονική στιγμή για να ε, προχωρήσει αυτό το θέμα. Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αναλάβω δέσμευση για προθεσμίες. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σιλοβίχη εκ μέρου των ε, φιλελεύθερων, παρακαλώ. Σίρι Όβιρ, λοιπόν. Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιο επίτροπε, στηρίζετε τη δημοκρατία και εγώ και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο μισός πληθυσμός ε, καταπιέζεται και είναι σε χειρότερη κατάσταση από ότι ο άλλος μισός πληθυσμός. Και αυτό επειδή τυχαίνει κάποιος να ανήκει στο γυναικείο φύλλο. Τα τελευταία 40 χρόνια, επαναλαμβάνω 40 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει χιλιόμετρα σελίδων αποφάσεων, οδηγιών, κατευθυντηρίων γραμμών, με δεσμευτική, με δεσμευτικό χαρακτήρα. Ακόμα όμως δεν έχουμε πετύχει την ισότητα. Είναι πολύ σημαντικό ότι και αν αποφασίζουμε, που όπως είπαμε έχουμε αποφασίσει πολλά, να τίθεται και σε εφαρμογή. Ρωτάω λοιπόν, αν δούμε τις διαφορές που υπάρχουν στους μισθούς, στις πληρωμές μεταξύ ανδρών και γυναικών, και εδώ δεν μιλάω για το 2007 που ήταν καλό, καλή χρονιά οικονομικά μιλώντας, θα δούμε ότι οι διαφορές στους μισθούς μεταξύ αντρών και γυναικών μάλλον έχουν αυξηθεί παρά μειωθεί στις χώρες μέλη. Εσείς τι θα κάνετε για να υποχρεώσετε τα κράτη-μέλη να τηρούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται για αυτό το θέμα στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνω... Ό,τι μπορώ. για να εφαρμοστεί υπάρχουσα νομοθεσία κυρίως το πρόβλημα παραμένει. Έχουν υπάρξει όμως βήματα προόδου τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Ιδιαίτερα αν εξετάσει κανείς το θέμα της διαφοράς αμοιβή ανδρών γυναικών παραμένει μια μεγάλη διαφορά αυτό το 17% σε ορισμένους τομείς αλλά τουλάχιστον σε σχέση με τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει υπάρξει πρόοδο στην Ευρώπη την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Πάντως τα προβλήματα παραμένουν, συμφωνώ μαζί σας. Οι διαφορές στην αμοιβή ανδρών γυναικών παραμένουν υψηλές και πρέπει να αντιμετωπίσουμε θετικά τις εμπειρίες ορισμένων χωρών όπως οι σκανδιναβικές χώρες όπου τα αποτελέσματα είναι καλύτερα και υπάρχουν πολλές γυναίκες σε υψηλά επίπεδα. μπορούν να υπάρξουν ε, προσπάθειες βοήθειας των γυναικών μέσω των αλλαγών στην οδηγία για την, για την ε, άδεια, τη γονική. Να βοηθήσουμε επίσης την καλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματικότητα. να προχωρήσουμε πάντα στην επιβολή του θέματος της αντιμετώπισης των διαφορών των φύλων σε όλες τις πολιτικές μας. Έχω μια συμπληρωματική ερώτηση. Αυτό το οποίο ήθελα να μάθω είναι αν οι αλλαγές, οι διαφορές μάλλον στις αμοιβέ ανδρών γυναικών μεγαλώνουν σε διάφορες χώρες. Εσείς μιλάτε για το 17% διαφορά. Στη δική μου χώρα είναι 33% αυτή η διαφορά. Εδώ και πέντε χρόνια ήταν 22%. Ποιο θα είναι το ποσοστό όταν κλείσει αυτή η οικονομική κρίση. Και η δική μου χώρα λοιπόν, αλλά και άλλες φοβάμαι, δεν στρέφουν την προσοχή τους σε αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών της Εσθονίας και ρωτάμε συνέχεια τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χώρες οι οποίες συνεχίζουν να παραβιάζουν τους κοινοτικού κανόνες. Αυτό το 33% στο οποίο αναφερθήκατε είναι το μεγαλύτερο ποσοστό διαφοράς το οποίο έχω ακούσει ποτέ. Και προφανώς θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε τέτοιου είδους ε, τεράστιες διαφορές. Να δούμε αν είναι αποτέλεσμα της κρίσης ή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και εκτός οικονομικής κρίσης. Όπως είπα πριν, υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να δει κανείς πίσω από τους μέσους όρους. Δεν γνωρίζω ακριβώς ποιο είναι το καθεστώς το οποίο ισχύει στη χώρα σας, αλλά υπόσχομαι να το εξετάσω και θα ζητήσω και από τις υπηρεσίες να με ενημερώσουν για τις πραγματικές αιτίες αυτής της κατάστασης, γιατί αυτό που μου είπατε είναι διπλάσιο από τον λεγόμενο μέσο όρο και είναι κάτι το οποίο καλεί να βρεθούν λύσεις αμέσως. Αν είναι κάτι το οποίο συνδέεται μόνο με τις διακρίσεις ανάμεσα στα φύλλα, τότε πολλά μένει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στις δύο ερωτήσεις τώρα από την Επιτροπή Πολιτισμού. Κύριος Παπα-Νικολάου. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Συζητήσαμε για τους... Εδώ κύριε, εδώ Επίτροπε. Μπροστά σας. Συζητήσαμε για την ανεργία στους νέους, για τη φτώχεια στους νέους. Ε, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις, ένας στους πέντε νέους τουλάχιστον αναφέρεται ότι ζει κοντά στα όρια της φτώχειας. Η ανεργία στους νέους είναι διπλάσια από ό,τι στο σύνολο των εργαζομένων. Ε, Παρ' όλα αυτά, όπως προκύπτει από πολλές ε, προσεγγίσεις, δηλαδή και από την προσέγγιση της τυπικής εκπαίδευσης αλλά και της μη τυπικής εκπαίδευσης, οι νέοι σήμερα έχουν περισσότερα προσόντα από ό,τι στο παρελθόν. Η κρίση ε, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την έβριση εργασία. Όταν τελικά όμω βρουν εργασία οι νέοι, συνήθω αυτή είναι κατώτερη των προσόντων που έχουν αποκτήσει και έτσι η επένδυση που έχουν κάνει στη γνώση δεν ανταποκρίνεται στι ανάγκε και στι προσδοκίε του. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που σας κάνω είναι, και τελευταίο βεβαίως σε αυτή τη φάση, πώς σκοπεύετε να διευκολύνετε και να ενισχύσετε τις δομές προκειμένου η μετάβαση από την γνώση στην αγορά εργασίας να είναι ευκολότερη και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των νέων. The uh, new skills for new jobs uh, νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα και θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης των εθνικών συστημάτων της αγοράς εργασία, όπως επίσης και των συστημάτων κατάρτισης για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στα οποία αναφερθήκατε, ιδιαίτερα η έλλειψη δεξιοτήτων ανάμεσα σε αυτούς που εγκαταλείπουν τα σχολεία και την εκπαίδευση γενικά. Η Εν πολλής είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως επίσης και κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών στο εσωτερικό των αγορών εργασίας και φτάνουμε σε υψηλότατα επίπεδα ανεργία των νέων που προκαλούν φτώχεια και μας υποχρεώνουν να δούμε τα πράγματα από πολύ κοντά γιατί τα προβλήματα αυτά σε μικρή ηλικία γίνονται διαρθρωτικά προβλήματα μακροπρόθεσμα και οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό. Και αυτό σημαίνει και πολύ υψηλότερο κόστος για την αντιμετώπιση τους. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά, τα δεδομένα αυτά και να χρησιμοποιήσουμε και την εμπειρογνωμοσύνη την οποία έχει συλλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα στοιχεία που θεωρούμε θετικά. παρόλα τα προβλήματα που αναφέρετε κι εσείς, οι νέοι που έχουν ε, κατά κοινή παραδοχή περισσότερα προσόντα από ό,τι στο παρελθόν, επαναλαμβάνω ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν σωστές προσβάσεις στην αγορά εργασία ανάλογα με τα προσόντα αυτά, παρά τα προβλήματα. Ο πιο πρόσφορος τρόπος για την πρώτη εργασιακή εμπειρία των νέων πλέον είναι τα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που και κατά τη διαδικασία αυτή, κατά την πρακτική άσκηση των νέων ανθρώπων, ε, οι νέοι, οι νέοι εργαζόμενοι που κάνουν την πρακτική άσκηση γίνονται ε, αντικείμενο εκμετάλλευση από του εργοδότε και τελικά καλούνται να καλύψουν ανάγκες πολύ περισσότερες από αυτές για τις οποίες η αποστολή των ε, προγραμμάτων αυτών υπάρχει. Σα ρωτώ, και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, στις περιπτώσεις αυτές όπου τα προγράμματα πρακτικής άσκησης ε, προσφέρονται και τελικά οδηγούν σε εκμετάλλευση των νέων ανθρώπων. Ε, θα κάνετε κάτι περισσότερο, θα έχουμε περισσότερους ελέγχους, θα λάβετε περισσότερα μέτρα. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα προγράμματα μαθητείας, αυτά τα προγράμματα τα προγράμματα μαθητείας στις διάφορες ε, χώρες ε, ήταν αν θέλετε ένας τρόπος για να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κρίση. Ε, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων εργασίας και οποτεδήποτε υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι νέοι σε θέσεις εργασίας, ε, δεν είναι προστατευμένοι, υφίστανται κακή μεταχείριση, δεν πληρώνονται, εσείς μάλιστα είπατε ότι μερικές φορές δεν πληρώνονται καθόλου. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους παρέμβασης. Το γεγονός βέβαια ότι υπάρχουν αυτά τα προγράμματα μαθητία, αυτό αποτελεί πρόοδο. Αυτό καθεαυτό. Τώρα, αν ε, καθοδόν παρουσιάζονται διάφορε ανομαλίε, βεβαίω αυτέ θα πρέπει να τι ερευνήσουμε και να δράσουμε αναλόγω. Τελευταία ερώτηση της Επιτροπής Πολιτισμού. Η Χόνιμπολ από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Θα ήθελα ε, κύριε Επίτροπε, να επιμείνω λιγάκι στο θέμα της ανεργίας των νέων. Τι μπορούμε να κάνουμε. Καταλαβαίνετε βέβαια από τον αριθμό των ερωτήσεων που ετέθησαν πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για μας ε, και πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμφίβολα ε, ένα κομμάτι του προβλήματος οφείλεται στα προσόντα. Θα συνεχίσω λιγάκι στην ερώτηση του κυρίου Παπα-Νικολάου. Δηλαδή, ιδιαίτερα σε σχέση με την ε, ανώτατη εκπαίδευση, όπου βλέπουμε να υπάρχουν απόφοιτοι που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους χωρίς προσόντα και τελικά σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να αποκτήσουν με άλλη μαθητεία και άλλα συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα. Πέστε μας, ποιες είναι οι λύσεις που ε, μπορούν να βρεθούν γιατί όλοι μας καταδικάζουμε και την ανεργία και τη φτώχεια, αλλά στη τελική ανάλυση αυτό που πρέπει να κάνουμε, όχι να καταδικάζουμε, να βρούμε μέτρα που θα βελτιώσουν την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορούμε τα προσόντα που αποκτούν οι νέοι να τα βελτιώσουμε, έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για τις θέσεις εργασίας, να υπάρχει αυτή η αντιστοιχία. Και Ίσως θα πρέπει ε, ένα στίγμα που υπάρχει σε κάποιες μορφές επαγγελματική εκπαίδευση. αυτό να πρέπει να καταπολεμηθεί, γιατί αυτό ξέρω ότι ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και είμαι σίγουρη ότι ισχύει και σε άλλες χώρες. Δεν είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι η επαγγελματική κατάρτιση πράγματι ε, μπορεί να ε, μεταφερθεί στα διάφορα επίπεδα που αφορούν τους νέους. Πρώτα απ' όλα, λέει ο Επίτροπος, να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα συνεχίσει να στηρίζει τις δραστηριότητες κατάρτισης συμπεριλαμβανομένου και του εξυγχρονισμού της επαγγελματικής κατάρτισης. Δεύτερο, θέλω να αναφέρω ε, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, που θα ασχοληθεί με τα προσόντα για τις θέσεις εργασίας και αυτή θα υποβάλει συστάσεις που θα αφορούν στο πώς ακριβώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πρωτοβουλία. Τον, την άνοιξη αυτού του έτους η Κομισιόν ε, θα εγκρίνει μία θα ανακοίνωση που κατ' ουσίαν θα προσφέρει κίνητρα για συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο μέλλον στον τομέα ε, της ε, επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι η περίφημη διαδικασία Κοπενχάγης όπως ονομάζεται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσει η Βελγική Προεδρία. Θα υπάρξει ανακοινοθέν σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Θα, υπάρξει ανακοινοθέν από αυτού. Ευχαριστώ. Έχουμε λίγο χρόνο για κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις και μια και τα πράγματα είναι αρκετά οργανωμένα, έχω ένα κατάλογο που να υπακούει πάντα στον κατάλογο Ντεχόντ και δίνω το λόγο στον κύριο Κλάρκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Άντορ. οι υπερβολικές ρυθμίσεις και οι υπερβολικές νομοθετικές ρυθμίσεις επηρεάζουν αρνητικά τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις τα καταφέρνουν γιατί έχουν πόρους, έχουν θα έλεγα αξιωματούχους που ασχολούνται με τη συμβατότητα των ε, τρόπων λειτουργία τους με την ευρωπαϊκή κοινότητα. Ε, κάποιες άλλες, ε, οι μικρότερες, έχουν πάρα πολλά προβλήματα και αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις και καταλαβαίνετε ότι οι μικρές επιχειρήσεις ε, αυτή τη στιγμή έχουν τις μισές θέσεις εργασίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί να αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα. Τι προγράμματα έχετε λοιπόν εσείς για τη μείωση του άχθους αυτούς που υφίστανται οι μικρές επιχειρήσεις. Ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι κρίσιμο σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, λέει ο κ. Σάντορ. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις αυτές. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σαν στόχο τη μείωση του αχρίαστου, του μη απαραίτητου διοικητικού βάρους και την απλούστευση των κανονισμών. Υπάρχει επίσης μια ομάδα υψηλού επίπεδου υπό την ηγεσία του κ. Στόιμπλ που προσπαθεί να μειώσει τη διοικητική γραφειοκρατία, την περιττή διοικητική γραφειοκρατία. Στον τομέα αυτό, επίσης, οι κοινωνικές ρυθμίσεις δεν είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, αυτού του είδους οι ρυθμίσεις επηρεάζουν πάρα πολλές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, που πολλές φορές κάνουν τη ζωή των επιχειρήσεων αυτών σχετικά δύσκολη. Αλλά οι κοινωνικές ρυθμίσεις, αυτές που ασχολούνται δηλαδή με την αγορά εργασίας, δεν είναι υπεύθυνε θα έλεγα για τα σημαντικά προβλήματα τα οποία μερικές φορές αντιποντοπίζουν οι επιχειρήσεις. Θα το εξετάσουμε, αλλά από τη δική μου πλευρά, από την πλευρά του δικού μου χαρτοφυλακίου οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες. Αλλά εγώ θα υποστηρίξω τις εργασίες της συγκεκριμένης αυτής ομάδας και θα ζητήσω την εφαρμογή των συμπερασμάτων τους. Αναφερθήκατε το, στις κοινωνικές ρυθμίσεις. Αυτό αφορά αυτούς που έχουν θέσεις απασχόλησης, αυτό το οποίο είπατε. Να επανέλθω προηγουμένως σε αυτό το οποίο αναφέρατε για την οδηγία για το χρόνο απασχόλησης, για το ωράριο εργασίας. Είπατε ότι δεν θα πιέσετε για να μειώσετε τα opt-out, τις εξαιρέσεις μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι, θα θέσετε, ότι δεν θα θέσετε μια ημερομηνία για να τερματιστούν τα λεγόμενα opt-out. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό από, με, νέο, τρόπο θα έλεγα. Αυτό το απαιτεί και η οδηγία για, το, για τα ωράρια εργασίας. Και θα πρέπει να τεθεί το θέμα σε ένα νέο πλαίσιο. Καταρχάς θα ήθελα να ακούσω τους κοινωνικούς εταίρους θα ήθελα να έχω συγκεκριμένα στοιχεία από μια μελέτη επιπτώσεων στον τομέα το συγκεκριμένο. Να πω επίσης ότι τα opt-outs δεν είναι απαραίτητα το καλύτερος τρόπος λύσης, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Από την άλλη, ε, εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να βάλω μία προθεσμία ή οποιαδήποτε μορφή προθεσμίας ε, για τέτοιου είδου συζητήσει σήμερα. Τελευταία Ευχαριστούμε. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Τατιάνα Στάνοκα από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Αξιότιμα υποψήφια επίτροπε. Εξαιτία τη κρίση, εδώ είμαι, εδώ είμαι, με βλέπετε. Κάποια κράτη-μέλη χρειάστηκε να ζητήσουν οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο μεταξύ η εφαρμογή των κοινωνικών μέτρων είναι πολύ αμφιλεγόμενη. Έχουν περιορίσει συντάξεις, για παράδειγμα, στη δικιά μου τη χώρα ή έχουν μειώσει τις ε, αποζημιώσεις ιατρικά έξοδα. Υπάρχουν ομάδες πιο ευάλωτες στις κοινωνίες μας που με την κρίση αυτή έχουν πληγεί ακόμα περισσότερο. Συμφωνείτε για το ότι ο κοινωνικός παράγοντας πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για την οικονομική στήριξη. Και αν ναι, πώς θα φροντίσετε για αυτό το θέμα. Η κοινωνική στήριξη δεν είναι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καταρχήν. Η αιρεσιμότητα αυτή από πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα έπρεπε να τίθεται σε εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια, την κρίση και τις φορολογικές πολιτικές που ανταποκρίνονται καλύτερα στην αντιμετώπιση της κρίσης. Δυστυχώς, οι συντάξεις μειώθηκαν, αλλά και θέσεις απασχόλησης σε μερικές περιπτώσεις. Οι υπάλληλοι και το δημόσιο τομέα βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση σε πολλές χώρες. Η κρίση είναι σκληρή και γι' αυτό ξεκίνησα στην εισαγωγή μου υπογραμμίζοντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε εξαιτία της κρίσης. πρέπει να αντιμετωπίσουμε καταρχήν τις αιτίε που οδήγησαν στην κρίση, να δούμε δηλαδή πάλι τη δημοσιονομική δομή και να παρθούν μέτρα για το μέλλον. Επί της παρούσης, ναι, πρέπει να βοηθούμε τις πιο ευάλωτες ομάδες, εκείνες που πλήττονται από τις περικοπές στις αμοιβές στις συντάξεις, και την ανεργία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Μεσματικό Ταμείο στηρίζει τέτοια προγράμματα και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και τέτοιου είδους προγράμματα βοήθειας προς αυτούς. Έχουμε λίγο ακόμα χρόνο για συμπληρωματικές ερωτήσεις. Εκ μέρους των φιλελεύθερων της Άλντε, η κυρία Νάντια Ήρς. Κύριε Επίτροπε, οι ερωτήσεις που αφορούν στους ε, θεσμούς, ε, συνδικάτα, επιχειρησιακά συμβούλια, σε αυτές απαντήσατε διεξοδικά. Όμως σε όλα τα άλλα θέματα που αφορούν εργαζόμενους όπως είναι οι νέοι ή οι ανάπηροι, Εκεί κρατηθήκατε στα πολύ γενικά. Εγώ όμως πιστεύω ότι τα προγράμματα και τα μέτρα που αφορούν ακριβώς αυτές τις ομάδες, πώς αυτές οι ομάδες θα επανέλθουν στην αγορά εργασίας, εκεί ακριβώς πρέπει κανείς να είναι χειροπιαστός και συγκεκριμένος για να τους στηρίξει. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, ο τομέας αυτός ε, που αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες να το πω καλύτερα, ε, για τα θέματα αυτά ε, ρωτήθηκε η κυρία Ρέντινγκ, μελλοντική σας συνάδελφος, αλλά εγώ σας ερωτώ και εσάς παρόλα αυτά. Θεωρείτε ότι πρέπει να είναι στοχευμένα τα μέτρα. Αναφέρετε τις ομάδες, παιδιά, αναπήρους, ομοφιλόφιλους, μετανάστες. Και αν ναι, αν συμφωνείτε για όλα αυτά, μήπως μπορείτε να προτείνετε και για τους ηλικιωμένους κάποια μέτρα. Όλα αυτά δηλαδή να είναι στοχευμένα. Ναι, πράγματι ε, πρέπει να συνεργαστώ με την κυρία Ρέντινγκ για όλους τους τομείς ε, στους οποίους εμφανίζονται φαινόμενα ε, διακρίσεων και όπου έχουν ληφθεί νομοθετικά μέτρα, έχουν εκπονηθεί νομοθετικά μέτρα. Σε όλους τους τομείς όπου τα κοινωνικά προβλήματα άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες που αναφέρατε, ανάπηρους ε, μετανάστες, πρέπει πράγματι να εκπονήσουμε στοχευμένα προγράμματα και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να καθορίσουν μόνα τους στόχους, έτσι ώστε να εφαρμόζονται πρακτικές ε, πρόσληψης ε, που προωθούν την αφομοίωση των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί βέβαια σε μία ή δύο ημέρες. Ε, αυτά τα θέματα πρέπει να ενταχθούν ε, στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 και πράγματι ε, αυτά τα θέματα θα είναι από τα βασικότερα που θα συζητηθούν την Άνοιξη. Να δούμε πώς μπορούμε να τα προβάλλουμε στην ατζέντα, στη μερίσια διάταξη των μακροπρόθεσμων θεμάτων. Θέλετε να επανέλθετε? Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι για σας αυτό είναι ένας ε, σημαντικός ε, τομέας στον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε πλήρως ε, στην κυρία Ρέντινγκ. Ο Επίτροπος, πρέπει να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να καλύψουμε όλα ε, τα στοιχεία που έχουν σχέση με την κατάρριξη των διακρίσεων. Αυτά τα καλύπτει η κυρία Ρέντινγκ. Όμως, παράλληλα, αυτά τα μέτρα ε, πρέπει να συνδεύονται και από κοινωνικά που είναι δικής μου αρμοδιότητας. Άρα δηλαδή αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο ερωτήσεις ακόμα και μετά ο Επίτροπος θα έχει πέντε λεπτά στη διάθεσή του, όπως προβλέπετε, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Επόμενη ερώτηση, η κυρία Όμεν Ράιτεν από το παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Άντορ, πολύ προσεκτικά άκουσα και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις και πραγματικά με ανοιχτό πνεύμα έχω να κάνω μια φιλική παρατήρηση. Σε όλες σχεδόν τις απαντήσεις σας χρησιμοποιείτε τη λέξη «εμείς», «we» στα αγγλικά. Εγώ θα προτιμούσα να λέγατε «εγώ» αντί για «εμείς». Και έρχομαι στα τέσσερα βασικά ζητήματα νομίζω. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα πλαίσιο για την υγεία είναι για τις Ευρωπαϊκές Ένωσης. Τι θα κάνετε με το πρώτο πρόγραμμα πλαίσιο λοιπόν, όπως ρώτησε και ο Στίβεν Χιούξ. Δεύτερον, κινητικότητα. Ο Τόμας Μάντ σας ρώτησε για αυτήν. Τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε για την 1η Μαΐου. Τρίτον, χρόνος εργασίας. Πρέπει να πω ότι οι αυτοξαιρέσεις, τα opt-out, δεν είναι ποτέ η λύση. Έχουμε την ανεργία, έχουμε κατευθυντήριες γραμμές και ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές στην Ευρώπη. Τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτή την τεράστια ανεργία 18% σχεδόν στην Ισπανία τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν έχουμε λύσεις. Πείτε μας λοιπόν συγκεκριμένα ποιο είναι το δικό σας πρόγραμμα. συνοψίσατε τα θέματα λίγο πολύ που συζητήθηκαν σήμερα. Το πρόγραμμά μου είναι να κοιτάξω το θέμα των στόχων της απασχόλησης και να φροντίσω να αποτελέσουν την προτεραιότητα στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να είναι πάνω-πάνω στην ημερήσια διάταξη. Χρειαζόμαστε την απασχόληση για την οικονομία. Πρέπει να βγούμε από την οικονομική κρίση και χρειαζόμαστε μία στρατηγική η οποία να λαμβάνει υπόψη της πολύ σοβαρά όλα αυτά τα θέματα και να προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις. Αυτή είναι η μερίσια διάταξη για την επόμενη περίοδο. Στην ακρόση σας μίλησα για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα. Είπα ήδη ότι θα ξαναδούμε το θέμα του χρόνου εργασίας και αναπόφευκτα θα ξαναγίνει συζήτηση μετά τον κοινωνικό διάλογο. Τα τελευταία χρόνια είχαμε μια νεοφιλελεύθερη επιρροή στην οικονομία της ε, κοινωνικής αγοράς. Τι θέλουμε από εσά. Από εσά θέλουμε να είσαστε ο Επίτροπος, ο οποίος νιώθει τα προβλήματά μας, τα προβλήματα των κοινωνιών μας και που αυτός ο συγκεκριμένος έρχεται με ένα πρόγραμμα πλαίσιο, ένα μάλλον πλαίσιο δράσης. Ο συγκεκριμένος Επίτροπος. Ναι, θα καταλήξω σε πρωτοβουλίες, αλλά προηγουμένως, λέει ο κύριος Σαντόρ, θα έχω χρησιμοποιήσει και τις αναλυτικές ε, ικανότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα λοιπόν θα έχω διάλογο με όλες τις πλευρές για τα διάφορα θέματα και μετά θα έρθω σε πρωτοβουλίες. Έχω σημειώσει όλα τα ζητήματα τα οποία μου θέσατε. Σας είπα ποια είναι η προσέγγιση μου, ποιος είναι ο προσανατολισμός μου και όσον αφορά τις πρακτικές και συγκεκριμένες λύσεις θα χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες και θα επανέλθω για διάλογο και θα ακούσω τις απόψεις σας για όλα τα θέματα που μου ζητήσατε τη γνώμη μου. Ευχαριστώ τελευταία ερώτηση από τους σοσιαλιστές Φρανσίσκο Ρώσα. Ε, Προήνση Αντερώσα, συγγνώμη. Προήνση Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, είσαστε ένας ήρεμος άνθρωπος σίγουρα και αυτό που θέλουμε εμείς να ακούσουμε από εσά στα τελευταία σας σχόλια είναι το κατά πόσο θα δώσετε τη μάχη για τις αρχές και τις πολιτικές που εσείς σήμερα μας υπογραμμίσατε εδώ. Γιατί στην Επιτροπή θα πρέπει να πάρετε θέση για τις διάφορες προτάσεις. Και εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι ο επίτροπο για τις Κοινωνικές Υποθέσεις θα αγωνιστεί για τους Ευρωπαίους. Θέλω κυρίω να σας ρωτήσω τη γνώμη σας για την κοινωνική πτυχή των εξωτερικών μας πολιτικών. Για τις προδιαγραφές που βάζει για την απασχόληση το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, για παράδειγμα ή το θέμα της εταιρικής ευθύνης. Ποια είναι η γνώμη σας για ρυθμίσεις σε αυτό το τομέα. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε απομονωμένοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις πιέσεις τις οποίες μας υποβάλλουν διεθνείς παράγοντες. Οπότε και αυτή η εξωτερική διάσταση είναι πολύ βασική. Εσείς θα τον δώσετε τον αγώνα, θα δώσετε τη μάχη. Ο κύριος Αντόρ, ναι, φυσικά θα τον δώσω αυτόν τον αγώνα. Πρόθεσή μου είναι όλα αυτά τα θέματα να τα πάρω πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά χρειάζομαι και τη δικιά σας τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Χωρίς τη στήριξη του Κοινοβουλίου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, εφαρμογή της τρέχουσας νομοθεσίας και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε νέες προτάσεις. Είναι προφανές ότι όταν μίλησα για συνεργασία μου με τους άλλους επιτρόπους, πρώτα συζήτηση, διάλογος, για να δούμε τα θέματα τα οικονομικά, της φτώχειας, των μεταναστών, των παιδιών, αλλά εννοείται ότι δεσμεύομαι υπέρ των καλύτερων λύσεων και θα φροντίσω να υπάρξει αυτή πρόοδο στα επόμενα χρόνια σε όλους αυτούς τους τομείς για τους οποίους μιλήσαμε σήμερα. Ευχαριστώ. Πολύ πολύ σύντομα για το θέμα της εταιρικής ευθύνης και τις προδιαγραφές ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας είναι στην ημερήσια διαταξή σας. Ναι, ψηλά μάλιστα στην ημερήσια διάταξη ακριβώς επειδή έχουν μια διεθνή διάσταση. Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι πολύ βασικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις έχουν τις δραστηριότητε τους σε πολλές διαφορετικές χώρες ή και υπήρους και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ηθικές πρακτικές. Αποτελεί και αυτό μέρος του χαρτοφυλακίου μου. Οπότε, εγώ θέλω να φροντίσω να πιέσω όλες τις χώρες να τηρούν τις προδιαγραφές του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, αν και περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Πρόεδρος, κύριε υποψήφια επίτροπε, απαντήσατε σε 40 ερωτήσεις από όλες τις πολιτικές ομάδες και τώρα έχετε στη διάθεσή σας 5 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 5 αυτά λεπτά ίσως και για να μας πείτε το πνεύμα της συνεργασίας που σκοπεύετε να έχετε με τα μέλη της Επιτροπής μας αυτής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικότερα εφόσον αναλάβετε τα καθήκοντά σας. Είναι αλήθεια ότι τα μέλη της Επιτροπής αυτής, τόσο παλιοί όσο και καινούργοι, νιώθουν συχνά μια απογοήτευση για τις διαπραγματεύσεις όταν είμαστε σε συναπόφαση, για παράδειγμα. Μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή, μεταξύ των δύο δηλαδή, προτιμάει το ένα σκέλος από το άλλο. Εσείς θα διορθώσετε αυτή την ε, στραβή, τουλάχιστον έτσι όπως την εισπράξαμε εμείς, κατάσταση. Έπειτα, πολλοί από τους ευρωβουλευτές εδώ λένε ότι στον κοινωνικό τομέα κατά βάθο υπάρχει νομοθεσία και ότι η δυσκολία μπορεί να ισχύει και αλλού. Αλλά σίγουρα εδώ, στον κοινωνικό τομέα, ότι η νομοθεσία αυτή που υπάρχει δεν εφαρμόζεται καλά από τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της την διαδικασία επί παραβάση. Μπορεί δηλαδή να πάει στο δικαστήριο μια χώρα μέλος εφόσον δεν εφαρμόζει ή δεν εφαρμόζει σωστά την κοινωτική νομοθεσία. Εσείς θα κοιτάξετε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα αυτό το μέσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε η νομοθεσία την οποία εγκρίνουμε εδώ με τόσο κόπο να τη βλέπουμε να γίνεται και πράξη στα κράτη-μέλη. Και όχι να απελπιζόμαστε στην Ευρώπη, αλλά αντίθετα να βελτιώνουμε την κατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών. Παρακαλώ λοιπόν ολοκληρώσετε και απαντήστε και σε αυτά τα δύο στοιχεία παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου προσφέρατε την ε, ευκαιρία να παρουσιάσω τη δική μου προσέγγιση, τις δικές μου απόψεις στην Επιτροπή σας. Νομίζω ότι η συζήτηση κατέδειξε ότι η κρίση είναι πράγματι, πράγματι πλήττει σκληρά την ευρωπαϊκή κοινωνία και αυτό αποτελεί μια δοκιμασία για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε όλοι από κοινού, να αναζητήσουμε λύσεις, διότι οι οικονομικές προκλήσεις θα παραμείνουν μεγάλες και τα βασικά θέματα, τα θέματα κλειδί του δικού μου του χαρτοφυλακίου, όλα αυτά επηρεάζονται από την κρίση. Κατά την άποψή μου, η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργαστούν στενά κατά τα επόμενα πέντε χρόνια και θεωρώ ότι η συζήτηση σήμερα ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική. Πρέπει λοιπόν να εκλειφθεί ως ε, το εναρκτήριο λάκτισμα. Τουλάχιστον αυτό ισχύει για εμένα. Πρέπει να βγούμε από την κρίση, οι άνθρωποι πρέπει να επανέλθουν στη δουλειά τους, ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, δομικές προκλήσεις που προέρχονται ε, από το περιβάλλον, στο περιβάλλον, από την ενέργεια. Υπάρχουν προκλήσεις επίσης και στην παιδεία και τέλος πρέπει να αναδιορθεί, αναδιαρθρωθεί γενικότερα η μακροοικονομική πολιτική. Αυτό το τελευταίο είναι και το πιο δύσκολο. Ορισμένες από τις ε, απαντήσεις που έδωσα στις ερωτήσεις ίσως να κρίθηκαν ιδιαίτερα γενικές. Όμως ε, θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα ε, είναι βασικό να συμφωνήσουμε, να καταλάβετε ότι δεσμεύομαι στην ιδέα της κοινωνικής Ευρώπης και είναι πολύ σημαντική η ημερήσια διάταξη, η ατζέντα του, για το 2020. Όσον αφορά τώρα τα θέματα που έθιξε που θίξατε εσείς κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι θεματοφύλακας της συνθήκης και οφείλει να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να ενισχύσει την κείμενη νομοθεσία. Εγώ τουλάχιστον θα το προσπαθήσω αυτό στο δικό μου τον τομέα, τον τομέα της απασχόλησης και των ε, κοινωνικών υποθέσεων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο ε, καλύπτει τώρα και νέα θέματα. Δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην ε, ένταξη των εργαζομένων ε, σε πράσινες θέσεις εργασίας, πολύ πιο σημαντικές αυτές από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα θεμελιώδη θέματα παραμένουν τα ίδια. Οφείλουμε να παραμείνουμε προσιλωμένοι στην πλήρη απασχόληση στην κοινωνική απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή και ελπίζω να κατάφερα να σας πείσω ότι εγώ προσωπικά ε, δεσμεύομαι για την ε, επίτευξη αυτών των στόχων. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ αυτή η τρίωρη ακρόαση. Ραντεβού στους συντονιστές για την αξιολόγηση της ακρόασης αυτής στις 8 στην αίθουσα 1 G2. 1G2.